ψήφιση του, του αιτήματος, ποιοι είναι υπέρ αυτών που ζήτησε το ΕΛΚ, ποιοι είναι κατά, ευχαριστώ. Επομένω, εγκρίνεται το αίτημα αυτό και η ψήφιση του σχεδίου κειμένου αναβάλλεται για την επόμενη ολομέλεια. Επομένω, εγκρίνεται η σε διάταξη τη Συνόδου και έχουμε παρακάτω κάποιε ανακοινώσει εκ μέρου του Πρόεδρου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ευχηθούμε το καλώ όρισε ει αυτήν την προσωπία της του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου. Επικεφαλή είναι ισότιμη με μέρη μου γέννη. Σήμερα μα επισκέπτονται. Είναι η δεύτερη αντιπρόεδρο του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου και είναι επικεφαλή τη αντιπροσωπεία για τη σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα δύο κοινοβούλια συνεργάζονται στενά. Επομένω, με μεγάλη μα χαρά θα σα έχουμε κοντά μα και με την ευκαιρία αυτή θα πρέπει να σα ευχαριστήσω διότι με προκαλέσατε να έρθω και να μιλήσω στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο όταν σε τρεις εβδομάδες θα έχετε σύνοδο. Δυστυχώς. Όμως δεν θα μπορέσω να παραστώ ίδιος αλλά θα στείλω ένα μήνυμα και πιστεύω ότι θα υπάρξει η ευκαιρία να τα ξαναπούμε Καλώς ορίσατε και πάλι. Το επόμενο θέμα πρόκειται για κάποιες δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής που αφορούν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο πρόκειται να συνεδριάσει. Πρώτα πρώτα καλώς ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Ζωζή Μανουέλ αλλά και ο Γκέγκο Λομπισγαρίδο, ο προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ μέρους του Συμβουλίου και θα δώσουμε ευθύς αμέσως το λόγο στον κύριε Υπουργό για να αρχίσει η συζήτηση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτούς τους μήνες που πέρασαν από τι αρχέ του 2010 είμαστε μάρτυρες μια πάρα πολύ έντονη δυναμική που στην Ευρωπαϊκή Ένωση. σοβούσε αυτής της πιο σοβαρής κρίσης που έχουμε γνωρίσει τα τελευταία 80 χρόνια. Ταυτόχρονα δε πρόκειται να τεθεί σε ισχύ μια νέα συνθήκη, συνθήκη της Λισαβόνας. Επίσης θα αρχίσει η λειτουργία κάποιων νέων θεσμικών οργάνων. Αλλά και ταυτόχρονα πρόκειται να έχουμε μια πάρα πολύ ε, εκτενή αναθεώρηση των οικονομικών μας συστημάτων. Και όλα αυτά γίνονται με κάποιο τρόπο, καμιά φορά άναρχο, άτακτο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικές οι προκλήσεις που βγαίνουν μπροστά μας. Να, για παράδειγμα, Έχουμε τώρα την αρρωγή προς την ελληνική οικονομία στην οποία ανταποκρίνεται η Ευρώπη με την συγκρότηση κάποιων νέων οργάνων και φορέων και μιας νέας οικονομικής πολιτικής προς όλες τις κατευθύνσεις και με όλες τους τις διαστάσεις. Καμιά φορά δεν μας αφήνει το δέντρο να δούμε το δάσος, αλλά έτσι κι αλλιώς πρέπει να δούμε πώς θα, τι θα σέψουμε αυτή την τόσο περίπλοκη οικονομία του 21ου αιώνα και αυτό πώς θα γίνει με προσέγγιση ευρωπαϊκή. Ακριβώς αυτό και κάναμε ανταποκρινόμενοι σε αυτήν την τόσο σοβαρή κρίση. Ήταν άμεση η αντίδραση του πώς κάποια κεφάλαια αντιστάθμισαν κάποια μεγάλα ελλείμματα τα οποία ανεφίσαν. Οπότε, αυτό το πρώτο κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε μια ε, μεγάλη αναθεώρηση της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και αυτό γίνεται με συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Είναι αυτό το οποίο έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία και θα κατεβάσει μια σχετική πρόταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να γίνει στη ζώνη του ευρώ, ένα συντονισμός, ούτως ώστε με αποφασιστικότητα να πάρουμε μια ξεκάθαρη στάση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τη σταθερότητα της Ευρωζώνης. Αυτό το Φεβρουάριο αποφασίστηκε, είναι μια δέσμευση πολιτική, ούτως ώστε να, να, να, να στεριώσει η σταθερότητα της Ευρωζώνης. Και στα πλαίσια όλων αυτών των δράσεων εντάσσεται και άλλη μία, δηλαδή το πώς θα βρούμε μια καινούργια στρατηγική καινουργια στρατηγικη αναπτυξη και ποιοτική απασχόλησης. Αυτό δε είναι το κεντρικό θέμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτή τη εβδομάδα. Πρόκειται για μια στρατηγική η οποία έχαράχθηκε και συνεχίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εκείνο το έγγραφο τη 3 η Μαρτίου που πρόκειται να μελετήσουν και να συζητήσουν στην Ιαρνή Σύνοδο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ακριβώ στα πλαίσια των στρατηγικών στόχων Αυτό μου διατύπωσε το εγγραφό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως την απασχόλησε. Την, επενδύσει σε έρευνα και ανάπτυξη, αλλά την ενέργεια και την αλλαγή του κλίματος, την εγκατάλειψη του σχολείου και του στήματος παιδείας, αλλά και την κατανόηση της φτώχειας. Επίσης, πρόκειται στο ε, Σύνοδο να συζητηθεί η διακυβέρνηση. Σε σχέση με το πού προσέχονται να υπάρχει δική της Λισαβόνας γύρω από τον άξονα της παρουσίας της πολιτικής ηγεσία του Συμβουλίου. Και επίση για το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει την εποπτεία του τι κάνουν τα κρατημέλη επί τη βάση των δεσμευσιών τους. Και αυτό πρόκειται να γίνει με στενή συνεργασία και έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των συναρμοδίων θεσμικών οργάνων τη Ένωση, αυτό είναι ο σκοπό τη συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και υπουργών. Καταπολέμηση τη αλλαγή του κλίματο, Πρωτοπορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνεχιστεί. Πρωτοπορία στη διεθνή σκηνή για την καταπολέμηση τη αλλαγή του κλίματο. Κάτι θα πρέπει να κάνουμε για να συνεχίσουμε να είμαστε πρωτοπόροι. Οπότε υπάρχει και μια πολιτική δέσμευση αυτό το οποίο ονομάζεται fast start. Ούτω ώστε να μπορεί να γίνει μια αποτίμηση από πλευρά του Συμβουλίου για το πώς προχωράμε για, αυτή μα την ε, δέσμευση, τι κάνουμε προ τι αντισομνές χώρες. Πώς καταπολύουμε την κλιματική αλλαγή και επίσης πρόκειται για πολιτική δέσμευση των ανεπτυγμένων χωρών. Συνεργασία των μεν με τις δε χώρες. Ούτως ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις αποφάσεις της Κανκούν. Άρα να συνεχίσουμε να είστε πρωτοπόροι και να κάνουμε το επόμενο βήμα μετά τα όσα συμφωνήθηκαν στην Κοπενχάγη. 27 στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνούμε βέβαια με τους στόχους της Κοπενχάγης και γι' αυτό και θέλουμε να έχουμε κάποιους στόχους, κάποιες, ε, κάποιες, κάποιες δεσμεύσεις, νομικά δεσμευτικές ε, πολιτικές υποσχέσεις για, για την Κανκούν του Μεξικού. Επομένως, αυτές είναι οι εξελίξεις τώρα. και όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κρίση που σοβεί στην Ελλάδα και για το πώς θα γίνει επαναχρηματοδότηση του δημοσίου χρέους της Ελλάδας και αναμφίβολα πρόκειται για μια πολιτική δέσμευση που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο αρχικών κρατών και κυβερνήσεων την 10η Φεβρουαρίου, ούτως ώστε να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε την Ευρωζώνη. Οπότε, εάν χρειάζεται να θεσπιστούν κάποια συγκεκριμένα μέτρα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την σταθερότητα, τότε θα ληφθούν αυτά τα μέτρα. Ακριβώς αυτό θα είναι το βασικό θέμα στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτή τη βδομάδα. Ευχαριστώ για τη δήλωσή σας κύριε Υπουργέ, εξ ονόματος του Συμβουλίου. Θα ήθελα να ζητήσω τώρα από τον πρόεδρο της Επιτροπής, κύριο Ζωζέ Μανουέλ Μπαρός, να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, είναι μια καλή και επίκαιρη στιγμή που συναντιόμαστε σήμερα μία μέρα πριν την σημαντική ανοιξιάτικη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας. Για να μπορέσουν αυτές οι προκλήσεις να ε, υλοποιήσουν είναι σημαντική η Συμβουλή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν λέγοντας αυτά να ευχαριστήσω και να συγχαρώ το Κοινοβούλιο για το ψήφισμά του σχετικά με την Ευρώπη του 2020 που υιοθέτησε στο Στρασβούργο πριν από δύο εβδομάδες με μια ευρεία υποστήριξη από όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω με την ίδια ευκαιρία την Ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου για την υποστήριξη που δίδει στην στρατηγική της Ευρώπης 2020. Η υποστήριξη αυτή εκφράστηκε σαφώς σε διάφορες συνθέσεις του Συμβουλίου των Υπουργών. Τώρα όμω έχουμε μπροστά μα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να πράξει δύο πράγματα. Ένα, να δείξει ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες της στιγμής και να δουλέψει και για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την Ευρώπη με συγκεκριμένους μακροπρόθεσμους στόχους. Η κρίση ε, σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές πιεστικές ανάγκες για τις κοινότητες, του εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Όπως γνωρίζουμε, σε εθνικό επίπεδο τα δημόσια οικονομικά υφίστανται άνευ πίεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά και την οικονομική, χρηματοοικονομική σταθερότητα και θα επανέλθω σε αυτά τα θέματα αργότερα. Η Ευρώπη, ωστόσο, δεν πρέπει να αγνοήσει την ανάγκη να δουλέψει τώρα για να επιτύχει μακροπρόθεσμε αλλαγέ. Γι' αυτό το λόγο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ασχοληθεί με δύο από του πιο σημαντικού μακροπρόθεσμου στόχου το οικονομικό μα μέλλον και την αλλαγή του κλίματο. Ήδη συζητήσαμε τη στρατηγική της Ευρώπης το 2020 στο Κοινοβούλιο. Η συνεισφορά και η δέσμευσή σας θα είναι απαραίτητες για να ολοκληρωθούν οι φιλόδοξες προθέσεις μας για μια έξυπνη, βιώσιμη και ε, πλήρη ανάπτυξη. Το ίδιο θα ε, λάβει υπόψη και το Συμβούλιο πολλά αναφέρθηκαν για το μέγεθος των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας και πρέπει να δείξουμε ότι έχουμε και συνοχή και όραμα. Και πρέπει να μπορέσουμε να περάσουμε αυτό στους ανθρώπους, να δείξουμε ότι η Ευρώπη κάνει τη διαφορά εκεί που μετράει. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό το Συμβούλιο να συμφωνήσει επί συγκεκριμένων στόχων αυτή την εβδομάδα. Οι στόχοι που έχει θέσει επιτάπητος η Επιτροπή επιλέγησαν προσεκτικά. Αντιμετωπίζουν την ανάγκη να αυξηθεί το επίπεδο απασχόληση, να δώσουμε περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και κοινωνία, να καλύψουμε τους στόχους ενέργειας και κλίματος του 2020, να βελτιώσουμε την εκπαιδευτική επίδοση και να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια. Αυτοί οι πέντε στόχοι ε, δείχνουν στόχους που μπορούν να με τους οποίους μπορούν να ταυτιστούν οι άνθρωποι και να δείξουν ότι η Ευρώπη παλεύει σε τομείς που είναι σημαντικοί και το ξέρουν όλοι δείχνει ότι έχουμε την πολιτική βούληση να αντιμετωπίσουμε σοβαρά και σκληρά προβλήματα. Βεβαίω θα πρέπει η στόχη αυτή να είναι επιτεύξιμη αλλά πρέπει να απαιτήσουν και μια επιπλέον προσπάθεια σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Μια αναγνώριση από τα κράτη-μέλη ότι χρειάζεται αλλαγή και θα προσπαθήσω να περάσω στα μέλη του Συμβουλίου αυτή την αίσθηση του επίγοντος για την σημερινή οικονομική κατάσταση της Ευρώπης και την ανάγκη μεταρρυθμίσεων ώστε να υπάρχει μια πιο βιώσιμη και ενωμένη οικονομία και κοινωνία στην Ευρώπη. Αυτό που είναι σημαντικό είναι τα μέτρα που θα λάβει κάθε κράτος μέλος για να, για να ενισχύσει το, ποσό οικονομικής, την το, το, το ποσοστό οικονομικής τους ε, Γεύθυνσης. Χρειαζόμαστε εθνικά μέτρα για την αντιμετώπιση των εθνικών ζητημάτων και με πλήρη τήρηση της επικουρικότητας, αλλά στο πλαίσιο ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου. Αν ένα μάθημα μπορούμε να ε, αντλήσουμε από αυτή την παγκόσμια κρίση είναι ότι όλοι είμαστε εξαρτημένοι από όλους. Δεν μπορούμε λοιπόν να δεχόμαστε ότι σε, ευρω... παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να υπάρχει κοινή ανταπόκριση αλλά σε εθνικό όχι. Χρειάζεται λοιπόν ένα κοινό πλαίσιο που θα πρέπει να ενισχύεται και να, ε, και να... Και να ε, από οικονομικά μέτρα με κάποιες, ε, με κάποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα δείχνουν ότι στο ευρωπαϊκό επίπεδο η Ευρώπη παρεμβαίνει σε κρίσιμους τομείς. Ψηφιακή ε, ατζέντα, καινοτομία, έρευνα βιομηχανική πολιτική και σε κάποιες περιπτώσεις βεβαίως θα βοηθήσει την επίτευξη στόχων σε εθνικό πλαίσιο, σε εθνικό επίπεδο. Προτείνουμε μια, ένα νέο ξεκίνημα χάρη στην ε, συνθήκη της Λισαβόνας μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια νέα ενισχυμένη προσέγγιση ε, συντονισμού και οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη δείχνοντας ε, συγκεκριμένους δυνατότητες στα κράτη-μέλη αντιμετώπιση των εθνικών στόχων αλλά με παρέμβαση, εντονότερη παρέμβαση της Ευρώπης ούτως ώστε να πάρει μπρος η οικονομία. Η αποδοχή της προσέγγισης αυτής θα είναι πραγματικά τεστ, ένα πραγματικό τεστ για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Με ενθαρρύνουν τα αποτελέσματα των άτυπο, του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ελπίζω ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πούν ναι όταν του ζητηθεί να ανταποκριθούν συλλογικά στις προκλήσεις αυτές. Σε ό,τι αφορά την αλλαγή του κλίματος γνωρίζω ότι το θέμα αυτό δεν μπορούμε να το αφήσουμε πίσω. Πρέπει να είναι στο πρώτο, πρώτο θέμα στην Ατζέντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι πρωτοπόρος. Έχουμε τους μόνους σαφείς μηχανισμούς μείωση των εκπομπών. Είμαστε οι πρώτοι δωρητές ενισχύσεων ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες σε θέματα κλίματος. Ας προχωρήσουμε λοιπόν, από, ας, αφήσουμε τις αναζητήσεις γιατί δεν πήγε καλά η Κοπεχάγη και ας προχωρήσουμε παραπέρα. Είναι σημαντικό να έχουμε σαφείς στόχους, συγκεκριμένες θέσεις. Γι' αυτό εξηγήσαμε, παρουσιάσαμε μια ανακοίνωση με τους στόχους ε, που θέλουμε να προωθήσουμε στις διεθνείς διαπραγματεύσει. Ταυτόχρονα η Επίτροπος ξεκίνησε τις διαβουλεύσεις με τους κύριους εταίρους. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια σαφή ε, προσπάθεια να προχωρήσουμε και να κλείσουμε συγκεκριμένες συμφωνίες μετά την Κοπενχάγη. Να κρατήσουμε το κύριο στην ημερήσια διάταξη, να κρατήσουμε ωστόσο σαφές ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο ε, με βάση μια διεθνή συμφωνία, όχι νωρίτερα. Και να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα κυρίως των ε, αναπτυσσομένων χωρών, δεσμευόμενοι λοιπόν ε, για την, αυτός δείχνει τη σημασία του fast start, του να χρηματοδοτήσουμε το fast start. Συνδέεται αυτό και με το στόχο της Ευρώπης του 2020 που περιλαμβάνει οικονομική, ε, οικονομικό εξυγχρονισμό και μεταρρυθμίσεις. Οι τομείς αυτής δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι προσβλέπουν για δράση στην ευρωπαϊκή πολιτική ηγεσία. Είμαι πεπισμένος ότι αν έχουμε την βούληση να είμαστε τολμηροί θα δείξουμε ότι η Ευρώπη έχει καθοριστική επίδραση στο μέλλον των πολιτών μας. Και με το πνεύμα αυτό θα παρουσιάσω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάποιες από τις βασικές προκλήσεις εν ώψη της, ομα... της συνάντησης της ομάδας των 20 που θα γίνει τον Ιούνιο στον Καναδά. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι κάποια από αυτά τα ζητήματα είναι ευρωπαϊκά αλλά θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν και σε παγκόσμιο επίπεδο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η οικονομική σταθερότητα και η χρηματοοικονομική κατάσταση στην Ελλάδα δεν είναι στην επίσημη μερίσια διάταξη αυτού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ωστόσο, για να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι δυνατό οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ιδίω αυτοί που μετέχουν στη ζώνη, στην Ευρωζώνη, να μην συζητήσουν το θέμα αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να σας δηλώσω τη θέση μας επ' αυτού. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια φάση διόρθωσης του υπερβολικού, ελλείμ, του υπερβολικού ελλείμματος. Η μείωση, σημαντική μείωση του ελλείμματος είναι κρίσιμη και η Ελλάδα έλαβε μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή. Ιδίω η Ελλάδα λαμβάνει μέτρα για την μείωση του ελλείμματός της φέτος κατά 4% σαν ποσοστό στο ΑΕΠ. Αυτή η δημοσιονομική προσπάθεια ευθυγραμμίζεται με την πορεία που έχει συστήσει η Επιτροπή και το Συμβούλιο, όπω αναγνώρισε στι 16 Μαρτίου και το ίδιο το Συμβούλιο. Βεβαίω, η, Ελλάδα, η δημοσιονομική προσπάθεια τη Ελλάδα πρέπει να συνεχιστεί, γιατί είναι ο μόνο τρόπο για να υπάρξει μόνιμη μείωση του κόστου τη χρηματοδότηση του χρέου ανταποκρινόμενη στην οικονομική και ε, χρηματοοικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, η άτυπη συνάντηση Υπουργού Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων στι 11 Φεβρουαρίου δήλωσε ότι τα κράτη-μέλη τη Ευρωζώνης θα αναλάβουν αποφασιστικό και συντον... αποφασιστική και συντονισμένη δράση, αν χρειαστεί, για την διασφάλιση τη οικονομική σταθερότητα στην ε, Ευρωζώνη συνολικά. Η Επιτροπή πιστεύει ότι είναι τώρα ενδεδειγμένο να δημιουργηθεί στο εσωτερικό της Ευρωζώνης ένα εργαλείο συντονισμένης δράσης που θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα σε περίπτωση που το την χρειαστεί. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι η δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού δεν θα περιέχει ε, αυτόματη ενεργοποίησή του. Η δημιουργία του μηχανισμού αυτού είναι και θέμα ευθύνης και αλληλεγγύης. Η αλληλεγγύη είναι αμφωτεροβαρή προσέγγιση. Η Ελλάδα καταβάλει μια οικονομική προσπάθεια στην προσπάθεια αυτή. Υποστηρίζοντα την προσπάθεια αυτή δεν βοηθάμε μόνο την Ελλάδα αλλά και την σταθερότητα τη ευρωζώνη συνολικά. Το πλαίσιο συντονισμένης δράσης θα πρέπει να θεωρηθεί ως δίκτυο ασφάλειας που θα χρησιμοποιηθεί μόνο όταν εξαντληθούν όλα τα άλλα μέτρα αποφυγής ε, ε, της κρίσης με πρώτα την ε, ε, εφαρμογή μέτρων πολιτική σε εθνικό επίπεδο. Πέραν των τεχνικών ε, διαστάσεων πρέπει η λύση να ενισχύει την συνοχή και την ενότητα της Ευρωζώνης και της διακυβέρνησής της. Η κοινότητα, ολόκληρη η κοινότητα χρειάζεται σταθερότητα. Η Ευρωζώνη είναι μια ζώνη σταθερότητας και είναι σημαντικό να ενισχυθεί περαιτέρω η δυνατότητά της να παρέχει σταθερότητα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για κάποια ζητήματα κυβερνητικά εργαλεία, αλλά αυτά τα εργαλεία πρέπει να ενσωματώνται σε ένα γιγαντιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι, είμαι πεποίθησή μου ότι η ανταπάντηση σε αυτή τη συγκεκριμένη πρόκληση θα αποτελέσει και ένα τεστ για τους Ευρωπαίους ηγέτες και για τη δέσμευσή τους προς μια οικονομική και νομισματική ένωση. Αυτό που διακυβεύεται είναι η ουσιαστική αρχή της, οικονομικής, της χρηματοοικονομικής σταθερότητας που βρίσκεται στο κέντρο της δημιουργίας του ευρώ. Και το ευρώ είναι ένα από τα πιο σημαντικά δημιουργήματα του ευρωπαϊκού εγχειρήματο και του ευρωπαϊκού οικοδομήματος μέχρι τώρα. Ελπίζω ότι το θέμα αυτό θα επιληθεί με πνεύμα ευθύνη και αλληλεγγύης. Αυτό είναι ο ευρωπαϊκό τρόπο για να πετύχουμε κάτι. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δήλωση αυτή, την εισαγωγική αυτή δήλωση. Και τώρα να ακούσουμε τις πολιτικές ομάδες. Ξεκινάμε με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τον Ζωζεφ Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η ομάδα του ΕΛΚ αναμένει από το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο να δηλώσει ξεκάθαρα την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, θέτοντας τον καθένα ενώπιον των ευθυνών του. Αυτό που προσδοκά η ομάδα του ΕΡΚ από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων είναι να ορίσουν ένα δρόμο για να βγει η Ευρώπη από την κρίση μέχρι πού θα μπορέσουν να συνεργαστούν και ποια είναι η κόκκινη γραμμή. Εκτιμά ότι η ανάκαμψη και η δημιουργία θέσεων εργασίας περνά από κοινέ δράσει με τα μέτρα που κάτι τέτοιο προποθέτει την επίτευξη τη χρησιμοποίηση τη καινοτομία, της εκπαίδευσης, της υποστήριξης στα ΜΜΕ, στις επιχειρήσεις, τη μάχη κατά τη ανεργία με τα αποτελέσματα που γνωρίζουμε. Υπενθυμίζω ότι τα κράτη-μέλη είχαν όλα προσυπογράψει το 2000 την προτεραιότητα στη στρατηγική της Λισαβόνας. Επειδή όμως δεν έδωσαν στους αυτούς τους τα μέτρα, επειδή δεν έβαλαν τους στόχους συγκεκριμένους, συγκεκριμένα, χάσαμε πολλά χρόνια. Και όλα όσα είπαμε έγιναν, αλλά εκτός της Ευρώπης. Η ομάδα μου λοιπόν περιμένει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πέρα των λόγων, να λάβουν σοβαρά υπόψη τους κοινού οικονομικούς στόχους βάσει των προτάσεων της Ευρώπης 2020 της Επιτροπής τροποποιημένη εκδοχή των οποίων θα παρουσιάσει το Κοινοβούλιο τον επόμενο Ιούνιο. Αλληλεγγύη. Πολύ, πολλά λέγονται εδώ και λίγε εβδομάδε για την ελληνική και που πραγματικά αποτελεί το Α και το Ω του ευρωπαϊκού οικοδομήματο. Από την δημιουργία τη ενιαία αγορά μέχρι την κοινή άμυνα περνώντα από το ευρώ. Η αλληλεγγύη αυτή ήταν ουσιαστική από το ξεκίνημα της χρηματοοικονομικής κρίσης. Δεν πρέπει να την στερήσουμε από τους, φίλους, από τους Έλληνες φίλους, όπως και από κάθε άλλη χώρα της Ένωσης που αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα. Αυτή την εβδομάδα πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε μια ευρωπαϊκή λύση στην κρίση αυτή. Και πρόκειται για, πρέπει να είναι μια κοινοτική λύση. Το επαναλαμβάνω, κοινοτική λύση. Αυτή είναι η λύση που πρέπει να λάβουμε υπόψη, σεβόμενοι τους ευρωπαϊκούς κανόνες και στα πλαίσια κοινοτικών μηχανισμών μηχανισμών χρηματοδότησης. Μόνο και μέσα στο πλαίσιο αυτό, αν θέλουμε, μπορούμε να εισάγουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πάντα όμως τηρώντας την κοινοτική, ε, τους κοινοτικούς κανόνες. Αυτό θα, προσπαθεί, θα επιτρέψει την λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Συστήματος. Αγαπητοί συνάδελφοι, από τη μια μεριά του νομίσματος είναι η αλληλεγγύη, από την άλλη είναι η ευθύνη. Η ευθύνη κάθε κράτους να τηρεί ειλικρινείς και σωστούς δημόσιους λογαριασμούς. Και τα κράτη που γνωρίζουν προβλήματα οικονομικά προς στιγμή πρέπει να κάνουν τις θυσίες, να δεχθούν τις μεταρρυθμίσεις που επιβάλλονται για να αλλάξει η κατάσταση όσο σκληρές και να είναι αυτές οι μεταρρυθμίσει. Με άλλα λόγια, η Ευρώπη πρέπει να είναι ελέγγυη προς την, Ευρώπη, προς την Ελλάδα, πρέπει να, την εξασφαλίσει ότι θα περάσει αυτή τη δύσκολη στιγμή. Αλλά βεβαίω και η Ελλάδα πρέπει στο εσωτερικό της να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσει που χρειάζονται βράχη και μέσο πρόθεσμα για να αξίζει αυτή την ελεγγύη. Και το πρότειναν χθε στο Κοινοβούλιο πρέπει να τα υλοποιήσουν. Αγαπη... Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η κρίση μα υποχρεώνει να αλλάξουμε. Η πρώτη αλλαγή αφορά στην Επιτροπή, που ζητώ να ασκήσει πλήρω και με δύναμη την ευθύνη που έχει ως θεματοφύλακα των συνθήκων. Η οι ρυθμίσεις του Συμφώνου Σταθερότητας πρέπει να εφαρμοστούν και αυτό πρέπει να το εξασφαλίσει η Επιτροπή και θα έχει την υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Δεύτερη αλλαγή αφορά την διακυβέρνηση των δημοσίων οικονομικών. Σε περιόδους ανάπτυξης ο καθένας θεωρεί ότι μπορεί να διασκεί φορολογική, δημοσιονομική και κοινωνική πολιτική χωρίς να ενδιαφέρεται για το κάνει ο άλλος. Σε περίπτωση κρίσης, σε περιόδους κρίσεων ωστόσο, αυτοί που έχουν δαπανήσει περισσότερα ζητούν την αλληλεγγύη αυτών που ήταν ας το πούμε πιο λογική μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Δεν το πιστεύω. Είναι καιρό στα κράτη-μέλη να, ε, να, να, ε, έχουν μεγαλύτερη σύγκληση των φορολογικών και ε, οικονομικών πολιτικών τους. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη κοινωτική διακριβένηση Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε. Αυτό ε, είναι απαιτεί και μεγαλύτερη αλλαγή. Αυτό είναι φυσικό. Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, σα καλώ να λάβετε σχετικέ πρωτοβουλίε. Γνωρίζετε, έχω μια κάποια εμπειρία πάντα σε περιόδους κρίσης προχωρά ο μηχανισμός και πραγματικά βιώνουμε αυτή τη στιγμή μία περίοδο κρίσης και έναντι των πολιτών και θεσμικά χρειαζόμαστε πολιτικό θάρρος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα εξ ονόματος ε, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο κύριος ε, Μάρτιν Σούλτς, ο πρόεδρος των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Σύνοδος πρέπει να ασχοληθεί με την κρίση στην Ελλάδα και πρόκειται να το κάνει. γράφει η International Herald Tribune σήμερα ότι η Ελλάδα υποσχέθηκε να κάνει τα μαθήματά της και να εξηγιάνει τον προϋπολογισμό της, τα δημοσιονομικά της. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, ζήτησαν από τους Έλληνες να το πράξουν αυτό ως προϋπόθεση για την παροχή αλληλεγγύης. Η Ελλάδα έτσι αναφέρεται στην εφημερίδα, ε, έδωσε τα αποτελέσματα που χρειαζόταν. Αυτός που τελικά δεν δίνει τίποτα είναι τα μέλη της Ευρωζώνης και πάνω απ' όλα η Γερμανία, η οποία αρνείται να κάνει το δικό της ε, τμήμα, το δικό της μέρος. Και έχει μίλησε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δικαίως για ένα δίκτυο ασφαλείας. Δεν είναι δυνατόν τα χρήματα του φορολογούμενου Τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Ιταλία, οποιαδήποτε χώρα να καταλήξουν στο Ταμείο της Ελλάδας. Όχι, δεν είναι αυτός ο στόχος. Το θέμα είναι η Ελλάδα να έχει την δυνατότητα να λάβει με τους ίδιους τόκους χρήματα από τις διεθνείς αγορές. Γιατί 2,5 μέχρι 3% είναι η φυσιολογική τόκη και χάρη λόγω ε, των κέντρων συνθήκων, πλέον η Ελλάδα καλείται να καταβάλει επιτόκιο 6%. Δηλαδή, τι γίνεται, τα χρήματα της εξυγίανσης που προσπαθεί να κάνει η Ελλάδα τελικά καταλήγουν στα, στις των κερδοσκόπων. Και μιλάμε για μια λαιλάτιση ουσιαστικά. Και είναι και παράλογο αυτό, είναι άτυχο, γιατί αν καθιερωθεί αυτό, αν αυτή η έλλειψη αλληλεγγύης οδηγήσει τέτοια κερδοσκοπία ενός κράτους της Ευρωζώνης, αν ε, τελικά αυτό καταστρέψει την εσωτερική αλληλεγγύη και τελικά αναγκαστεί να παρέμβει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όχι η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη, τότε η κερδοσκοπία θα χτυπήσει τη Βρετανία, την Ιταλία, την Ισπανία. Θα είναι, αν θέλετε, μόνο ένα πρώτο βήμα η Ελλάδα. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε αλληλεγγύη προς την Ελλάδα. Γι' αυτό η αλληλεγγύη προς την Ελλάδα Και αυτό κυρίω θα πρέπει να το εξηγήσουμε στη Γερμανίδα Κακελάριο αποτελεί μια πράξη οικονομικής λογικής. Δεν πρόκειται για παροχή βοήθεια έτσι, ανεφαντελάγματος. Δεν μπορούμε λοιπόν ε, να απαλλάξουμε τον κύριο Μπαρόσο από τις ευθύνε του. Λέγοντα ότι αν λύσει αυτά το, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υποβάλει προτάσει για το πώ στο ιστορικό τη Ευρωπαϊκής ε, της Ευρωζώνης θα επανέλθει η σταθερότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω υπέβαλε καλέ προτάσει και θεωρώ ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να ανταποκριθεί στις προτάσει αυτέ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Αυτό δεν σημαίνει, ε, δεν συνεπάγεται, δεν ε, συμπεριλαμβάνει χρήση του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Και γιατί. Γιατί είμαστε σε θέση να επιλύσουμε το θέμα αυτό, το πρόβλημα αυτό στο ιστορικό τη Ευρωζώνη. Και μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός το γεγονός ότι η Άγγελα Μέρκελ θέλει να εμπλακεί το Διεθνές, Ευρωπαϊκό, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ε, η γερμανική Bundestag, η γερμανική τράπεζα, ε, λέει ότι η συμβολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την επίλυση διαρθρωτικών ε, προβλημάτων σε ό,τι αφορά δηλαδή, τη χρηματοδότηση των ε, ε, δημοσιονομικών ελλημάτων ή των τραπεζών με την νομισματική του εντολή δεν συνάδει. Δηλαδή δεν συνάδει αυτή η εντολή. Αυτό το λέει η Γερμανική Τράπεζα και Τράπεζα. Και αναφέρεται Αντιθέτω, ε, από, την από την Γερμανία τα καγκελάρια ότι θα πρέπει να λύσει το πρόβλημα το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Δεν είναι σωστό τρόπο αυτό. Χρειάζεται να στείλουμε ένα μήνυμα προ τι διεθνεί αγορέ. Ότι κερδοσκοπείτε όσο θέλετε. Δεν πρόκειται να αποσταθεροποιήσετε την Ευρωζώνη. Αυτό το μήνυμα χρειαζόμαστε. Μόνο τότε θα σταματήσουν οι κερδοσκοπίε. Και γιατί κερδοσκοπίε μιλάμε. Αυτό να το δούμε στα swaps. Είναι σαφές. Τα credit default swaps. Κλείνω δηλαδή μία ασφάλεια, ασφάλιση ότι θα καεί το σπίτι του γείτονα. Και όταν καεί το, σπίτι του γείτονα θα, θα εισπράξω το ποσό της ασφάλισης. Αν έχω συμφέρον να καεί το σπίτι του γείτονα, αλλά τι λέει ο Φλόριαν άναψε φωτιά στα σπίτια των άλλων. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεται αυτό στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν η αλληλεγγύη προ την Ελλάδα αποτελεί πράξη σταθεροποίηση τη Ευρωζώνη. Να αποφασίσουμε τι θέλουμε σε τελική ανάλυση. Θέλουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη ή θέλουμε να τα αφήσουμε τα πράγματα στην τύχη του. Εγώ δεν θέλω να πω ότι συμφωνώ, αλλά αναφέρεται από το Financial Times της Γερμανίας. Δεν είναι σοσιαλιστικό, ξέρετε, ε, το έντυπο αυτό. Σας παρακαλώ να ακούσετε με προσοχή τι αναφέρθηκε ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, αναφέρεται στο Financial Times της Γερμανίας, όπου υπάρχει ευρωπαϊκή ανάγκη αντίθετη με το γερμανικό ε, λαϊκισμό. Και πρέπει να διαλέξουμε. Ας αποφασίσουμε να κάνουμε αυτό που επιτάσσει η ευρωπαϊκή ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο Σούλτς. Ε- Και τώρα εξ ονόματος ε, των φιλελευθέρων. Ο κύριος Χι Βερχοφστάτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι το, το συμπέρασμα μπορούμε όλοι να αντλήσουμε ΕΛΚ, πράσινοι, σοσιαλιστές, φιλελεύθεροι και νομίζω και όλοι οι άλλοι. Ίσως και οι ευρωσκεπτικιστές. Είναι ότι τώρα θα πρέπει κύριε Πρόεδρε να βρούμε πώς θα υπάρξει κάποια ξεκάθαρη θέση του Συμβουλίου της Ευρώπης γιατί πρόκειται τώρα για δύο εβδομάδες που έχουμε κλείσει ε, όπου εκτός των θεσμικών Οργάνω γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση για το τι μπορούμε να κάνουμε για την Ελλάδα και για την Ευρωζώνη. Αυτό είναι χωρίς προηγούμενο, γιατί έχουμε δύο εβδομάδες που δεν αναλαμβάνουμε αποφάσεις απλώς, ε, διαφωνούμε, τσακωνόμαστε για το τι, τι μέτρα θα πάρουμε. Θα πάρουμε το, το α ή το αντίθετο του α. Τη μια μέρα στην άλλη. Και πρόεδρε, εκτό από αυτό δημιουργείται η εντύπωση ότι μέσα σε τέσσερι μέρε είχαμε κάποια μέλη του Συμβουλίου τα οποία δεν κάνανε τίποτα για το ευρωπαϊκό όραμα. Κάνανε πιο κακό από όσο μια τετραετία όλοι μαζί οι ευρωκευτικιστές. Αυτό αυτή είναι η εντύπωση έχω. Επομένω, ο μόνο τρόπο για να αλλάξει κάτι τέτοιο είναι να έχουμε μια αποφασιστική στάση και απόφαση από τη βάση πρόταση τη Κομισιόν. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενο που σήμερα μα το είπε ο πρώτο Μπαρόζο ότι πρόκειται να κατεβάσει πρόταση στο Συμβούλιο για μια λύση, μια λύση ακριβώς όπως είπε ο κ. Ντούλου, το οποίο συμφωνώ ότι θα πρέπει να πρόκειται για λύση που να είναι ευρωπαϊκή, κοινοτική και να μην είναι αυτό που λέμε εδώ και μήνε, ότι δηλαδή θα πρέπει να πάρουμε τα χρήματα τη τσέπη των φορολογουμένων για να τα δώσουμε, γιατί δεν πρόκειται περί αυτού. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να υπάρχει ένα ε, όργανο, ένα μέσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο ώστε να συρρυκνωθούν τα επιτόκια των, ε, του δανεισμού της Ελλάδας, των ομολόγων. Και αυτό δεν είναι θέμα μόνο αριθμιστή για την Ελλάδα, πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι χρειάζεται ρευστότητα και αξιοπιστία. Και δύο πράγματα χρειάζονται όσον αφορά για τα, τα, τα επιτόκια. Αυτά τα δύο που σας είπα. Έχει η Ευρώπη δυνατότητα και στην αξιοπιστία και στην ρευστότητα. Αυτό θα πρέπει να γίνει και ούτε ένα ευρώ ένας φορολογούμενος να μην ε, δοθεί στην Ελλάδα. Και αυτό όμως είναι πάρα πολύ αναγκαίο γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το, το, το, το spread είναι 3%, 3, κάτι το, το, το, το ομόλογο το, το γερμανικό και τώρα είναι 6,50 σήμερα το ελληνικό. Άρα το spread είναι 3,5, 3,5 μονάδες βάση. Επομένως ο μόνος λόγος αυτό να αρθεί είναι να κάνουμε αυτό το οποίο χρειάζεται Δηλαδή να βρεθεί ένα μέσο ευρωπαϊκό. Άλλος λόγος όμως να το κάνουμε αυτό είναι ότι ε, θα καταβάλουν, είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν οι Έλληνες κάποιες προσπάθειες που να βγουν σε, σε, κάτι καλό. Γιατί εάν δεν βρεθεί μια ευρωπαϊκή λύση, εάν δεν κατέβουν τα επιτόκια, τότε όλες αυτές οι προσπάθειες θα, θα πέσουν στο κενό, όλα αυτά θα πάνε στις αγορές των κεφαλαίων. Αν δεν υπάρξει μια αποφαστική στάση του συμβουλίο. Προσπάθειες ε, εξοικονόμηση δαπανών και ποιος θα κερδίσει οι κεφαλαίοι αγορές, οι κερδοσκόποι, εκείνοι οι οποίοι θα μπορέσουν να αποσπάσουν ακόμα καλύτερα επιτόκια. Γι' αυτό θα πρέπει να πανεύει η Ευρώπη, ούτως ώστε η εξυγίνηση της ε, οικονομίας της Ελλάδας να χρησιμεύσει. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι στηρίζουμε και όλο το Κοινοβούλιο θα πρέπει τώρα να στηρίξει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επομένω, ήρθε η ώρα να σταματήσουν οι κουβέντε στο Συμβούλιο και ήρθε η ώρα να εγκρίνουν την πρόταση τη Κομισιόν. Σα ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρεμπέκα Χάραμ, εξ ονόματο των Πρασίνων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω εν συντομία πόσο σύντομα όταν ε, αντιμετώπισαν ε, προβλήματα οι τράπεζες στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, πόσο σύντομα λοιπόν σε μία νύχτα σε πολλές περιπτώσεις αποφασίστηκε να συνδράμουμε στις τράπεζες αυτές και αυτό αποτελεί συζητάμε ακόμα σήμερα μάλλον δεν συζητάμε ούτε καν σήμερα τους όρους ε, για τη βοήθεια αυτά, για τη βοήθεια αυτή. Δεν τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά. Και αν το συνειδητοποιήσουμε λοιπόν αυτό και αντιληφθούμε ότι η ελληνική κρίση, η κρίση της Ελλάδας, η κρίση του ευρώ ουσιαστικά αποτελεί ευρωπαϊκή κρίση και θα πρέπει συζητιέται εδώ και εβδομάδες ολόκληρες, μήνες, χωρίς οι Ευρωπαίοι πολίτες να βρουν το θάρρος να κάνουν αυτά που χρειάζονται. Ουσιαστικά πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι ντροπιαστικό και ως Γερμανίδα και ως Γερμανίδα βουλευτής εδώ στο Κοινοβούλιο ντρέπομαι για την κυβέρνησή μου. Γιατί διαβάζουμε σήμερα ότι λαμβάνει η χώρα στις Βρυξέλλες η Ειδική Σύνοδος μόνο υπό τον όρο ότι θα αποφασιστεί για την Ελλάδα αυτό που θέλει η κυρία Μέρκελ προκειμένου να φύγει ε, στεφανωμένη με Δάφνες ε, ως νικήτρια για να επιστρέψει στη, στο Βερολίνο, αυτό πραγματικά το βρίσκω όνειδος. Και εκεί θα μας έχουν νικήσει οι φυλάδες, αν θέλετε. Και θα πρέπει, κύριε Λάγκα, να το σκεφτούμε αυτό και ιδιαίτερα στην γερμανική αντιπροσωπεία, αν αυτό επιτρέπεται, αν ε, θέλουμε αλληλεγγύη ή δεν θέλουμε αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό, δηλαδή, συγγνώμη, εξαρτάται από δημοσκοπήσεις ε, που κάνει ε, ένα γερμανικό κόμμα για τις εκλογές σε ένα κρατήδιο. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί απαράδεκτο λαϊκισμό και είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν ορίζεται σήμερα ότι στην σύνοδο της Πέμπτης και της Παρασκευής θα αποφασίσουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων τι θέλουν να κάνουν, τι θα, μέτρα θα πάρουν για την κρίση στην Ελλάδα. Επειδή παρακολούθησα τόσο στενά την ε, συζήτηση που γίνεται στη Γερμανία και βρέθηκα και στην Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα, θα ήθελα να πω ότι οι πολίτες ε, στη χώρα μου και η αλληλεγγύη για την ε, παροχή σωστών ε, δανείων ε, προς την Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει μόνο όταν δεν πρόκειται για μονόδρομο. Τα θέματα αυτά τα οποία συζήτησα στην Ελλάδα μου κατέδειξαν ότι οι πολίτες στην Ελλάδα έχουν τώρα την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα καλύτερο κράτος. Αυτό το κράτος θα πρέπει να αξιοποιήσει την κρίση για να πραγματοποιήσει πραγματικές μεταρρυθμίσεις και σε κανέναν, ε, κανέναν δεν ωφελούμε αν δεν υποστηρίξουμε την διαδικασία αυτή, αν δεν στηρίξουμε τον κύριο Παπανδρέου στην ε, διαδικασία αυτή. Κυρίες και κύριοι, επειδή έχω ζήσει πάρα πολύ στενά λαϊκισμό στη Γερμανία, θα ήθελα να σας δώσω και μία άλλη οπτική. Η δική μας ανάλυση είναι η εξής, ότι το ευρώ μπορεί να έχει ουσία ως κοινό νόμισμα αν οι Ευρωπαίοι ε, κινηθούν προς μία σύγκληση της ε, οικονομικής τους πολιτικής, γιατί ο ανταγωνισμός είναι αυτός που οδηγεί σε δυσκολίες. Στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σήμερα και έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Και πολλά θα πρέπει, θα κληθούμε να εξηγήσουμε στους πολίτες για την ανάγκη της ε, ενοποίησης. Το κάναμε αυτό και όταν συζητήσαμε ε, το Σύνταγμα, τη Συνταγματική Συνθήκη. Χαιρόμαστε που πλέον έχει τεθεί σε εφαρμογή η συνθήκη της ε, Λισαβόνα. και στην, πρόχη, στην πρώτη μάχη να μα κερδίσουν οι φυλάδε, ο κίτρινο τύπος, η κυρία Μέρκελ θα έκανε μεγάλο λάθος αν δεν πατήσει φρένο γιατί το βασικό είναι η ανάγκη της ε, οικονομικής ενοποίησης. Αυτό θα πρέπει να συζητηθεί. Θα πρέπει να παρουσιάσουμε διαφανή και πιστικά επιχειρήματα προς τους πολίτες μας. Όχι να αφήσουμε την Bill, την εφημερίδα, να τα εξηγήσει όλα. Ιδάλλως, άμα γυρίσει τιμένη η κυρία Μέρκελ, θα γράψει δηλαδή η Bill ότι να καταργήσουμε το ευρώ και τι θα κάνουμε στην περίπτωση αυτή. Δεν έχουμε ακόμα, έχουμε ακόμα περιθώριο επιλογής, δεν έχει περάσει ο χρόνος ο κρίσιμος και νομίζω ότι ελπίζω ο κ. Σαρκοζή να είναι πιο λογικός από την κυρία Μέρκελ. Ευχαριστώ για την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, ο κ. Καμίνσκι. Κύριε Πρόεδρε, στην Ολομέλεια έχουμε αυτή τη στιγμή μια συζήτηση για την Ελλάδα, έστω και αν δεν είναι επίσημα στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θέλω να εκφράσω το σεβασμό προς την ελληνική κυβέρνηση. Ε, γίνονται διαδηλώσεις στους δρόμους. Έχει εξεγερθεί το ίδιο το εκλογικό σώμα της Ελλάδος για την αλληλεγγύη, την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη ως στόχο προς το συμφέρον της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης η κυβέρνηση να λαμβάνει σκληρά μέτρα και λυπούμε που βλέπω ότι δεν είναι όλοι οι ευρωπαίοι ηγέτες έτοιμοι να αντισταθούν στον λαϊκισμό. Πιστεύω ότι η Ευρώπη χρειάζεται αλληλεγγύη, η Ελλάδα χρειάζεται αλληλεγγύη γιατί η Ευρώπη είναι χτισμένη πάνω στην αλληλεγγύη. Βεβαίω δεν πρέπει να επιτρέπουμε σε οποιονδήποτε πολιτικό, σε οποιαδήποτε χώρα να αντιμετωπίζει την οικονομική πολιτική ω εάν ήταν ένα είδος καροτσάκι σε σούπερ μάρκετ. Αυτό κάνουμε στην Ελλάδα. Στο μέλλον θα πρέπει να υπάρξουν σκληροί κανόνες για τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να επιδιώκουν ορθολογικές, σωστές, εύλογες οικονομικές πολιτικές. Μια οικονομική πολιτική που δεν στηρίζεται σε ορθές βάσεις δεν θα επιτύχει και λυπούμε που λέω ότι σήμερα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η ιδεολογία και η πολιτική ε, πάνω από την οικονομία. Αυτό είναι λυπηρό η Ευρώπη, πιστεύω, μπήκε στο ευρώ πολύ νωρί, υπερβολικά νωρί. Επειδή ωστόσο δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην πολιτική παρά στην οικονομία, επιτρέπηκε να ενταχθεί στο ευρώ η Ελλάδα. Ελπίζω ότι η Επιτροπή σήμερα θα λειτουργήσει ως θεματοφύλακας και της Ευρωπαϊκής Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής κοινή Λογικής. Χρειαζόμαστε αλληλεγγύη, χρειαζόμαστε όμως και λογική. Κύριε Πρόεδρε, με δεδομένη την σημερινή οικονομική κρίση. Δεν θα έπρεπε να προσπαθούμε να δώσουμε ένα φάρμακο που θα επιδεινώσει την κρίση. Μεγαλύτερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη ρυθμιστική προσέγγιση. Αυτά δεν θα βοηθήσουν να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε την υιοθέτηση την, την, την επιβολή των γραφημοκρατών στην κοινή αγορά. Θα πρέπει να τηρούμε και να σεβόμαστε τις διαφορές μεταξύ πολιτιστικών, ιστορικών και λοιπόν διαφορών που υπάρχουν μεταξύ κρατών μελών. Ναι λοιπόν στην ελληνική προς την Ελλάδα και θα ήθελα να εκφράσω εκ νέου το βαθύ σεβασμό μου προς την ελληνική κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, ο κύριος Λότρο Μπίσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σπάνια συμφωνώ και με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, αλλά όταν ζητούν και οι δύο αλληλεγγύοι προς την Ελλάδα και μιλούν για, προειδοποιούν μάλλον για την επανεθνικοποίηση, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί τους, γιατί σωστά μιλούν ο κύριος ε, Μπαρόσο ανέφερε στο Στρασβούργο πως θα πρέπει να απαγορευτούν οι κερδοσκοπίες στην αγορά και η αυξημένη, ο αυξημένος διχασμός στις κοινωνίες, στις ε, ευρωπαϊκές κοινωνίες δεν μπορεί να παραβλεφθεί. Προκύπτουν και ανακύπτουν ε, πολλά σημαντικά ερωτήματα τα οποία δεν είναι στην ημερήσια διάταξη των αρχηγών των κυβερνήσεων και θα πρέπει να συζητηθούν φυσικά η συζήτηση για την Ευρώπη του 2020 αναφέρεται. Όπως ξέρετε η ομάδα μου δεν είναι ενθουσιασμένη για τη στρατηγική αυτή γιατί ειλικρινά είναι η, αυτή, αυτός ο ανταγωνισμός ο αποτυχημένος που προκάλεσε την κρίση. Θέλουμε μια Ευρώπη η οποία θα θέτει τα κοινωνικά, την κοινωνική ανάγκη πάνω από τον ανταγωνισμό και προς αυτήν την κατεύθυνση η Ευρώπη και η σχετική της στρατηγική το 2020 απέχει παρασάγκας. Αλλά όταν ε, κοιτάζουμε τους στόχους αυτούς σε ό,τι αφορά για παράδειγμα του, την απασχόληση, την έρευνα και την εκπαίδευση, τη φτώχεια. Τι γίνεται ε, με τη στατική του 2020, το έτος της καταπολέμησης της ένδυας. Ελπίζω αυτή η στάση να μην επικρατήσει στην πλειονότητα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο Μπίσκι. Και τώρα η κυρία Νίκη Τζαβέλα. Κυρίες και κύριοι, η πατρίδα μου η Ελλάδα έχει πολλά κοινά σημεία με την Καλιφόρνια. Έχουμε πολύ ωραίο κλίμα, το περιουσιακό μας στοιχείο είναι η γη μας. Καήκαν τα δάση μας όπως καήκαν και τα δάση στην Καλιφόρνια. Κάναν Ολυμπιακούς αγώνες όπως κάναμε και εμείς καταλήξαμε να έχουμε τα ίδια προβλήματα με την καλιφόρνια. διαρωτώ με κύριε πρόεδρε εάν η καλιφόρνια είχε πρόβλημα δανεισμού θα αφήνονταν από την κεντρική κυβέρνηση των ηπα έρμεο των κερδοσκόπων. It's the economy, yes, it is. Το καταλαβαίνω και γι' αυτό είπα αυτό που είπα προηγουμένως. Έλληνε η κεντρική κυβέρνηση, τον είπα. Έχουμε ή δεν έχουμε κεντρική κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα η οποία αντιστοιχεί στο 2% της ευρωπαϊκής οικονομίας έχει δημιουργήσει τόσο μεγάλο πρόβλημα στο ευρώ, έχει πριονίσει τη συνοχή του ευρώ και απειλεί την ενότητα της Ένωσης. Είναι σαφές λοιπόν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα crash test στις αντοχές του ευρωνομίσματος αλλά κυρίως και στις προθέσεις των ηγεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να το υπερασπιστούμε. Αν κάνουμε μία αναδρομή τι έχουμε επιτύχει τριάντα χρόνια πριν ήμουν νεαρή υπάλληλο μικρή υπάλληλο του υπουργείου εργασία και εκπαιδευόμουν εδώ στι βρυξέλλε για την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. έχουμε επιτύχει την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά έχουμε επιτύχει το ευρώ. δεν νομίζω ότι επιτύχαμε τίποτα άλλο κοινό γι' αυτό με βλέπετε και στους ευρωσκεπτικιστές. ελπίζω λοιπόν αύριο να αποδείξουμε ότι πράγματι έχουμε αποδείξει μια σύμπνοια και κάτι κοινό κύριε πρόεδρε. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο πρόεδρος και ο επόμενος ε, αγορητής είναι ο Ζόλταν Μπάλτσο για τους ε, αδεσμεύτους ανεξαρτήτους. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο και πρέπει να σας πω ότι κάποιοι από τους προλαλήσαντες μας ε, μίλησαν για το ποια θα πρέπει να είναι πιο δόκιμη λύση στο ελληνικό πρόβλημα. Όλοι τέλος πάντων σε αυτό αναφέρθηκαν. Κύριε ε, Μπαράσο, τι έγινε με την ε, ημερήσια διάταξη της συνάντησης κορυφής. Γιατί είστε τόσο υποκριτές που δεν έχετε βάλει το θέμα στη μέση διάταξη. Ισχύει το ότι μόνο η Ελλάδα βρίσκεται σε δυσκολία γιατί και η Ουγγαρία πέρσι βρισκόταν στο χείλο του γκρεμού γιατί γίνανε πάρα πολύ σημαντικά λάθη από την κυβέρνηση. Είχαν γίνει κάποιε λαδροχέ με τον ε, ε, προπολογισμό και αυτό έχει πάρα πολλέ σοβαρέ συνέπειε. Επομένω, θα πρέπει από το credit crunch να αντιλήσουμε κάποιες, ε, κάποια μαθήματα, κάποια συμπεράσματα και να δράσουμε αναλόγω. Επομένω, αυτό είναι το πραγματικό μάθημα που πρέπει να αντιληφθούμε τα τελευταία 20 χρόνια από τότε που κατέρευσε το τείχο του Βερολίνου. Από τότε γινόμαστε μάρτυρε τη κατάρρευση τη Wall Street. Επομένω, και κοιτάξτε τι γίνεται σε παγκόσμια κλίμακα γιατί νομίζω ότι αυτό το σύστημα έχει γίνει κάτι σαν κράτος εν κράτη στην ε, διεθνή οικονομία. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος και τώρα το λόγο έχει ε, ε, το τμήμα των Αγωγητών που αφορούν τις πολιτικές και πρώτης είναι ο Γκαρφία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Εσείς ξέρετε περισσότερο από όλους πόσο θέλει να βοηθήσει το δικό μου κόμμα την επιτυχία της πανική Προεδρία. Κάντε διόρθωση πορεία. Και κάντε αυτό το οποίο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Προεδρία σημαίνει να βρεθεί μια λύση για την Ελλάδα. Αυτό το είπαν όλοι και να μην επαναλάβω και εγώ τα ίδια. Επομένω, να έχει κανεί το τιμόνι τη ε, Προεδρία είναι το να βρεθούν κάποιε εναλλακτικέ επενδύσει, να μην καθυστερούμε τι εξελίξει. Θα πρέπει το νωρίτερο δυνατόν να εγκληθεί. Να εγκριθεί μια, μια δέσμη αποφάσεων για εποπτεία χρηματοοικονομική και να μην ε, είναι συντηρητικό το, το Συμβούλιο, που είναι πιο συντηρητικό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέση με την πρότασή τη. Και είναι ακόμα πιο συντηρητικό από την ε, έκθεση Λαροζιέλ. Ε, το Κοινοβουλίο μα πρόκειται προ την Προεδρία ε, να δώσει το πράσινο φω για μια, συμφωνία. Συμφωνία για την εποπτεία. Και αυτό συνοψίζεται στο σύνθημα περισσότερη υποπτία, περισσότερη Ευρώπη. Εμεί πάντοτε αυτά τα, τα, πρεσβεύουμε και πιστεύω ότι και, και όσοι θέλουν το καλό τη Ευρώπη να ακούσουν αυτή τη φωνή και όχι άλλε. Να συμφωνήσουν με το Κοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε περισσότερη δημοσιονομική πειθαρχία και αναβαθμίζοντα την πειθαρχία σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε κάποιε φρέσκε ιδέε, ούτω ώστε να δρούμε προληπτικά και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η αναθεώρηση των 14 ε, προγραμμάτων σταθερότητας ήταν τελικά μια ενέργεια γραφειοκρατική διότι απουσιάζει οποιαδήποτε ε, ιδέα προληπτικής φύσης. Επομένως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ανταγωνισμός των οικονομιών γιατί χωρίς ε, πλούτο δεν λένε τίποτα οι δημόσιοι λογαριασμοί. Επομένως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το εξωτερικό ισοζύγιο. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες κυρώσεις ώστε να υπάρχει μια δεσμευτική πλευρά σε αυτό το σύμφωνο. Επίσης μας μιλήσατε για την διακυβέρνηση, τα, τα, είπαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωση, επομένως ξέρετε ότι είχαμε το άρθρο 121 και το 136 της ε, συνθήκης της ε, Λισαβόνας και αυτά θα επικαλεστεί τώρα η Προεδρία και θα πρέπει να δούμε τι άλλο χρειάζεται. Ό,τι χρειάζεται να μα το πείτε, θα σα βοηθήσουμε. Αλλά για να σα ε, βοηθήσουμε θα πρέπει να ξέρουμε τι πρεσβεύετε. Τι πρεσβεύετε και τι επιθυμείτε. Γιατί ξέρετε, τα κούφια λόγια δεν πιάνουν εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Το λόγο είχε ο κύριος Χιούγκς. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύουμε ότι τα σχέδια συμπεράσματων του Συμβουλίου που είδαμε όλοι ε, μπορεί να αποτελέσουν πραγματικό κίνδυνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα συμπεράσματα μιλούν για μια επίκαιρη έξοδο από μέτρα υποστήριξη. Τι σημαίνει αυτό. Το είδαμε στα συμπεράσματα του ΕΚΟΦΗΝ χθε. Θέλουν να φύγουν από το 2010 τα μέτρα υποστήριξη αγορά. Το Συμβούλιο του Δεκέμβριου μίλησε για την ανάγκη να επανέλθουμε στο, στα κριτήρια του Συμφώνου Σταθερότητα μέχρι το τέλο του 2013 για όλα τα κράτη-μέλη. Πιστεύουμε ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι απελπιστικά αισιόδοξο. Εάν ακολουθήσουμε την προσέγγιση αυτή, ε, την επιστροφή δηλαδή στα κριτήρια του Συμφώνου Σταθερότητας, ε, θα οδηγηθούμε σε τεράστιες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, σε αύξηση της ενεργείας, σε ε, μία περίοδο ε, αργής ανάπτυξης που θα, οδηγήσει σε μείωση των οικονομικών ε, δυνατοτήτων για πολλά χρόνια. Θα είναι συνταγή καταστροφής. Χρειαζόμαστε μια έξυπνη ισορροπία μεταξύ υπεύθυνη φορολογικής πολιτικής αφενός και συνεχιζόμενης υποστήριξης αγορά από την άλλη. Χρειαζόμαστε μια ε, βιώσιμη και μόνιμη στρατηγική εξόδου από την κρίση. Το Δανικό Ινστιτούτο Εργασία έδωσε κάποια στοιχεία και είπε ότι οι συμφωνίε εξόδου από την κρίση ε, που έχουν συμφωνήσει 20 κράτη-μέλη με την Επιτροπή θα απαιτήσουν 4,5, θα, χωρίς τα μέτρα αυτά, 4,5 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει, θα προσθεθούν στις τάξεις των ανέργων. Αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Άρα χρειάζεται να υπάρξει ένα μορατόριο δύο ετών για, την, ε, για διακοπή των μέτρων εξόδου από την κρίση, των μέτρων υποστήριξης ε, της αγοράς εργασίας. Ελπίζω, θα ήλπιζαν ήταν παρόν ο κ. Μπαρόζο, θα του ζητήσω να θα του έλεγα ότι δεν μα πειράζει όταν παίρνει τι ιδέε αν έπαιρνε τις ιδέε μας και τι παρουσίαζε σαν πρότασή του στο Συμβούλιο αύριο. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Εκ, για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Το Συμβούλιο θα συναντηθεί αύριο για να συζητήσει το μέλλον μια Ευρώπη που αντιμετωπίζει τεράστιε προκλήσει. Αντί αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε την οικονομική κρίση, την κρίση στην, στην αγορά της εργασίας, την κλιματική κρίση. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει μια πραγματική οικονομική ανάκαμψη για να πάρει μπρος η Ευρώπη. Φοβούμαι ωστόσο ότι οι προτάσει του Συμβουλίου και τη Επιτροπή για τη διακυβέρνηση τη Ευρώπη θα είναι υπερβολικά ασαφεί και θα βοηθήσουν την επίτευξη των στόχων. Αν εφαρμοστεί ω έχει η πρόταση για την Ευρώπη το 2020, θα είναι ό,τι ήταν η στρατηγική της Λισαβόνας, μια αποτυχία. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει ε, κα, ε, ε ενώπιος τις προκλήσεις αυτές. Με κάποιες προτάσεις. Πρώτον, η μέθοδος ανοιχτού συντονισμού δεν λειτουργεί, πρέπει να εγκαταλειφθεί. Αντίθετα, πρέπει να υιοθετηθούν δεσμευτικοί στόχοι που θα επιθέτει η Επιτροπή βάσει των, στό, των δυνατοτήτων που προσφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας. Αν ένα κράτος μέλος δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις εν ώψη της ε, στρατηγικής 2020, δεν θα πρέπει να δαπανούμε ε, περαιτέρω οικονομικά κονδύλια. Ναι λοιπόν στην ελεγγύη αλλά και στη διαφάνεια. Τρίτον, η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύει τι αιτήσει εκθέσει με συστάσεις πολιτική στο Κοινοβούλιο πριν συζητηθούν στο Συμβούλιο. Πρέπει να δημιουργηθεί μια ανοιχτή διαδικασία που θα επιτρέπει πολί, πολίτες να εμπλακούν πραγματικά. Ω Ευρωπαίοι πολιτικοί πρέπει πάντα να προσπαθούμε να θέτουμε του πολίτε στο κέντρο τη πολιτική μέσα. κάνουμε λοιπόν την πραγματικότητα πολιτική και ας ε, ενσωματώσουμε, ας κάνουμε την Επιτροπή έναν τίγρη που να διαθέτει δόλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσίλε έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να συζητήσουμε όχι μόνο την περίπτωση της Ελλάδας, αλλά και το σύνολο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Κοιτώντας τι γίνεται με την στρατηγική της του 2020, θεωρώ ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνει έμφαση όχι τόσο στην οικονομική συνοχή και θα πρέπει αυτό να το θεωρήσουμε στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών ε, προοπτικών για το 2014 μέχρι το 2020 το στοιχείο της οικονομικής συνοχής είναι απόλυτα απαραίτητο και κρίσιμο. Με άλλα λόγια, αυτό τι σημαίνει ότι μέχρι τότε θα πρέπει να έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της συνοχής, γιατί μετά το 2020 θα είναι ακόμα πιο μεγάλο το χάσμα από ότι τώρα. Αυτό θέλουμε. Αυτό αποτελεί την ε, ιδέα της αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να το εξετάσει αυτό με πιο πολύ σοβαρότητα και να δώσει συγκεκριμένους οικονομικούς στόχους. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα ο κύριος Χατζηγεωργίου. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, έχουμε ασχοληθεί νομίζω αρκετά και δίκαια με το θέμα της Ελλάδας. Εγώ θέλω να θίξω ένα ζήτημα που αφορά και άλλες χώρες. Ο κύριος Σούλτς έχει πει ότι σήμερα το επιτόκιο στην Ευρώπη είναι 2-3%. Εγώ θέλω να σας πω ότι στην Κύπρο το επιτόκιο σήμερα είναι 6%. Είναι γονατισμένες οι τράπεζες πάνω σε αυτό το επίπεδο και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει αυτή την εικόνα. Θεωρούμε ότι το Συμβούλιο πρέπει να εργαστεί και προς την κατεύθυνση του μέλλοντος για να μην δούμε άλλα κράτη να μπαίνουν σε αυτόν τον κυκαιώνα που έχει μπει η Ελλάδα. Θέλω να βάλω δύο εισηγήσεις. Δώσαμε δισεκατομμύρια, κυρία Πρόεδρε, στις τράπεζες με στόχο να κυλήσει η οικονομία. Έχω μια εισήγηση. Δεν θα ήταν καλύτερα το κράτος να έδιδε αυτά τα λεφτά ως επιτόκιο για το δάνειο πρώτης κατοικία, εφόσον ο καταναλωτή πήγαινε στο ταμείο για να πληρώσει τη δόση του. Και μια δεύτερη εισήγηση. Δεν θα μπορούσαμε να δούμε την επιβολή φόρων στις μεγάλες συναλλαγές τις διασυνοριακές μεταξύ των κρατών. Και μια φράση για το ένα λεπτό κυρία Πρόεδρε, με συγχωρείτε θέλω να το πω. Το ένα λεπτό δεν επιτρέπει σε κάποιον να στοιχειοθετήσει την άποψή του. Στο τέλος τέλος είναι και ένας εξευτελισμός να καταντάς να λέει συνθήματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταλαβαίνω ότι σε ένα λεπτό δεν μπορείτε να διατυπώσετε όλες σας τις απόψεις. Ένα λεπτό για τον κύριο Μπορκέτσι όμως. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι απλό να διαχειριστεί κανείς την Ευρωζώνη. Κάθε μέρα αντιλαμβανόμαστε ποιοι είναι οι κίνδυνοι, τους οποίους μας περιέγραψαν πολλοί συνάδελφοι, αλλά οι ηγετικέ προσωπικότητες στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Υπουργοί Οικονομικών, ακόμα δεν έχουν εξευρυλίσει. Ίσως να είναι ε, αδύνατη αυτή η αποστολή και όλα εξαρτώνται από το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο και τι θα αποφανθεί. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τις οικονομικές προδιαγραφές έχει επιμείνει συγκεκριμένα να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ασχολόμαστε υπερβολικά με τις τράπεζες, αλλά τι γίνεται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη δική μου χώρα, στην Ιταλία, τα διευθυντικά ταμεία σε κάποιες περιφέρειες χρησιμοποιούνται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά μόνο το 2% απορροφάται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, θα πρέπει να ασχοληθεί πολύ πιο εντατικά με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος, ο κύριος Λάγκεν. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω έναν έπαινο προς την Ελλάδα γιατί μόνο σκληρά μεταρρυθμιστικά μέτρα της Ελλάδας θα λύσουν το πρόβλημα της Ελλάδας. Όλα τα υπόλοιπα που προτάθηκαν είναι κατά των ευρωπαϊκών συνθήκων και αναμένω και από τον Πρόεδρο της Επιτροπής αλλά και από το Κοινοβούλιο αυτό να τηρήσουν τις συνθήκες και να μην υποβάλουν προτάσεις αντίθετες προς τη σύμβαση. Στον συνάδελφο Σούλτς να πω ότι φωνάζοντας δεν αντικαθιστά την εμπειρογνωμοσύνη. Δεν είναι οι κερδοσκόποι αυτοί που προκάλεσαν τα προβλήματα της Ελλάδας, αλλά οι ιστορικοί κανόνες, η απροθυμία των κρατών μελών να τηρήσουν το σύμφωνο, το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης και η Γερμανία και η Γαλλία ήταν οι κακοί, οι κακές χώρες όταν έδωσαν το παράδειγμα αν δεν αλλάξουμε τους κανόνες, αν δεν υπάρχει η προθυμία αυτή να τηρήσουν τα κρατημέλη τους παλιούς κανόνες, εκεί ξεκινούν τα προβλήματα. Και τώρα να λέμε ότι φταίνε οι κερδοσκόποι, γιατί ξέρετε το λιγότερο, το μικρότερο ποσοστό του ενός τρίτου των ε, χρέων της Ελλάδας προήλθαν από τους κερδοσκόπους. Άρα πρόκειται για δικαιολογία. Όσο δεν είμαστε σε θέση και οι Υπουργοί Οικονομικών είναι οι κακοί. Όσο δεν είμαστε σε θέση να τηρήσουμε τους κανόνες που έχουμε θέσει, θα αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Αυτό είναι η λύση. Η λύση δεν είναι να επιτιθέμεθα σε έναν μόνο ηγέτη μιας ευρωπαϊκής χώρας ή στο συνταγματικό δικαστήριο της χώρας μας. λέει Ο κύριος Βόμποντα, 1,5 λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι σαφές και συνάδελφε για το ακούσαμε ότι η Ελλάδα φυσικά θα πρέπει να κάνει τα δικά της ε, μαθήματα, αλλά είπαμε και με σαφήνεια ότι πρέπει να υπάρξει και αλληλεγγύη, αλληλεγγύη η οποία θα βοηθήσει η Ελλάδα να καταφέρει να κάνει τα μαθήματά της. Και όταν κοιτάμε τα ποσοστά την κερδοσκοπία που δεν ευθύνεται για την κρίση στην Ελλάδα, αλλά για τα τεράστια χρέη που τώρα θα πρέπει να αναλάβει η Ελλάδα. Αυτό είναι το καθοριστικό, κύριε Λάμε. Κάτι που είπαν οι Financial Times ότι αυτή είναι η διαφορά του κυρίου Κόλ και της κυρίας Μέρκελ. Ο κύριος Κόλ θα έλεγε να επιλύσουμε το πρόβλημα εδώ και τώρα μαζί με την Ελλάδα. Και η κυρία Μέρκελ τι κάνει, προσπαθεί να ξεφύγει. Λέει, α, να δούμε τι λένε οι συνθήκες, τι λέει το συνταγματικό δικαστήριο. Αυτή είναι η πολιτική διαφορά. Δηλαδή, τι κάνουμε, κοιτάμε την πολιτική ενοποίηση, την ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κοιτάμε τι γίνεται στην πατρίδα μας. Κανείς δεν ζήτησε να χαθούν αυτά τα χρήματα. Αλλά όταν δρούμε μόνο λαϊκιστικά και δεν σκεφτόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η κακοφωνία προκαλείται. Ή μια άλλη εφημερίδα, η Εφατσέτη, η οποία ανέφερε ότι κάθε μέρα προβάλλεται και υποβάλλεται ξεχωριστή πρόταση. Δεν δίνονται οι σωστές απαντήσεις και αυτό είναι απαράδεκτο γιατί ναι, δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Χρειαζόμαστε τα μέτρα αυτά στην Ελλάδα, τα οποία θα πρέπει να είναι σκληρά, αλλά θα πρέπει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε την παρουσίαση τέτοιων προβλημάτων και αυτό μπορεί να συμβεί άσχετα με το αν θα προκύψει Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, μόνο μέσω ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Και αυτό περιμένω από τη Σύνοδο. Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για να διαμορφώσουμε καλύτερα το μέλλον από ό,τι είναι τώρα διαμορφωμένο. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Χολ για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η Σύνοδος της Άνοιξης κανονικά θα έπρεπε να ασχοληθεί με το θέμα της ενέργειας. Αν υπήρχε υπάρξει μια συμφωνία στην Κοπεχάγη θα συζητούσαμε ήδη τι τεχνικές συνέπειες τη μείωση των εκπομπών κατά 30%. Αυτό πρέπει να το κάνουμε παρά τα αυτά. Πρώτον, διότι οι φιλοδοξίες που επιτεύχθηκαν στην, άνοιξη, στο, στην Σύνοδο κορυφή της άνοιξη του 7 μιλούν για πολύ μεγαλύτερη μείωση, απαιτούν πολύ μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών. Την περασμένη εβδομάδα ο εκτελεστικός διευθυντής ε, της εξαιρετικά επιφυλακτική διεθνού επιτροπή ενέργεια, δήλωσε στου ευρωβουλευτέ ότι η εικόνα του, της ενέργειας του IAA για το 2009 προβλέπει μείωση 3% της γενικής παραγωγής ενέργειας και ότι το 30% είναι σωστός στόχος. Επίσης, η μείωση του στόχου κατά ε, του, της χρήσης ενέργειας το 2050 σημαίνει απαιτεί να μειώσουμε τουλάχιστον κατά 30% την χρήση άθρακα στην ενέργεια το 2020. Για να μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε και μια αποτελεσματική οικονομία ε, και δημιουργία θέσει εργασία, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την προσέγγιση τη μείωση τη χρήση ε, άνθρακα στην ενέργεια. Θα έπρεπε λοιπόν να υποστηρίξουμε σαν ότι είναι αναγκαίες συνθήκες για να προχωρήσουμε στον στόχο του 30%. Επίσης, το Συμβουλίο θα έπρεπε να γνωρίσει ότι ο φθηνότερο τρόπος για να επιτευχθεί αυτή η περικοπή είναι με την αποτελεσματικότητα της ενέργεια, ιδιαίτερα δε με δεσμευτικού στόχου ε, αποτελεσματικότητα ενέργεια. Η Ένωση πρέπει να περάσει ένα σαφέ μήνυμα στην σύνοδο αυτή όπως έκαναν και στη σύνοδο του 2007. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζημάνσκι έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, αντί να μιλάμε για την εφαρμογή της Ατζέντα του 2020, θα μιλήσω για κάτι άλλο, κάτι που μπορούμε να επηρεάσουμε στην ουσία να προστατεύσουμε την εσωτερική αγορά από τον προστατευτισμό, να κάνουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία ευκολότερη για τους επιχειρηματίες, να έχουμε καλύτερη νομοθεσία, κάτι που είναι ευθύνη του Κοινοβουλίου. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να θα προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις αν υπάρξει πίεση από την παγκόσμια οικονομία. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε στα κράτη-μέλη την μέγιστη δυνατή ελευθερία στο, στις φορολογικές ε, εταιρικέ και κοινωνικές ρυθμίσεις που υιοθετούν. Η ελευθερία είναι ε, η απάντηση στην κρίση, όχι το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Ευχαριστώ. Η κυρία Βότμαν Κόλ για δύο λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ε, υπάρχει ακόμα τέτοια λύση κατεπίκουσα για την Ελλάδα και αυτό δεν αποτελεί ακόμα πρόβλημα γιατί ακόμα και ο Έλληνας ε, Πρωθυπουργό είπε ότι η Ελλάδα θέλει να λύσει μόνη της τα προβλήματά της και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ακολουθήσουμε το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης και αυτό είναι αλληλεγγύη. Ωστόσο έχουμε ένα πρόβλημα. Στην παρούσα φάση το ευρώ πέφτει κατακόρυφα και αυτό, αυτό το προκαλούν οι ανοιχτές συζητήσεις μεταξύ των ε, πρωτευουσών, αν δεν μπορέσουμε να βρούμε μία λύση. Ελπίζω λοιπόν αυτό το πρόβλημα να επιληθεί αύριο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ένα δίκτυο ασφαλείας, ε, όπου θα πρέπει να συνεργάζονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ελπίζω, κύριε Πρόεδρε, να κοιτάξουμε περαιτέρω αύριο τα αίτια της ε, κρίσης και επίσης τις λύσεις βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τα προληπτικά μέτρα του προγράμματος σταθερότητας και ανάπτυξης και η καινούργια στρατηγική του 2020 μπορεί να στεφτεί μόνο με επιτυχία, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, μόνο αν υπάρχει πραγματικά ευρωπαϊκή διακυβέρνηση στη βαρύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεργαστούν μόνο τα κράτη-μέλη στη Σύνοδο, αλλά και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ό,τι αρμοδιότητες της δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας, προκειμένου πραγματικά να ενεργήσει και να προβεί σε συγκεκριμένε πράξεις, Γιατί μόνο με την ελευθερία δεν θα καταφέρουμε τίποτα, όπω είπατε. Ελπίζω αύριο, κυρία Πρόεδρε, πριν από την έναρξη της Συνόδου, να γίνει αυτή η συνειδητοποίηση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κρίση και στην Ολλανδία με μια καλή, στεναρή στρατηγική το 2020 μετά την Κοπεχάγη. Ο κύριος Χουντής, για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από δηλώσεις αξιωματούχων αλλά και από δημοσιεύματα του τύπου το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται ω το πιο επικρατέστερο σενάριο διάσωσης εντός εισαγωγικών της ελληνικής οικονομίας, μια σύμπραξη χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Διεθνές νομισματικό ταμείο. Ε, Ενδεχομένω προ τα εκεί και η κυρία Μέρκελ. Θα, θα ήθελα να σα πω, κύριε συνάδελφε, ότι αυτό είναι το χειρότερο, το πιο αντικοινωνικό σενάριο τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρωζώνη. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα τέτοιο ενδεχόμενο παραδιάζει την κοινοτική νομιμότητα και το λέω για αυτούς που την υπερασπίζονται κατά τα άλλα καθώς σε καμία συνθήκη, σε κανένα νομικό κείμενο δεν αναφέρεται καμία τέτοια παρέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή άλλου διεθνούς οργανισμού σε αυτές τις διαδικασίες. Ταυτόχρονα δημιουργείται ένα προηγούμενο πολιτικό και νομικό καθώς αυστηροποιεί το σύμφωνο σταθερότητας και εισάγει από το παράθυρο της ΗΠΑ στην Ευρωζώνη. Όσον αφορά την Ελλάδα, μια τέτοια επιλογή θα εντείνει στο έπακρο τα αντεργατικά και αντικοινωνικά μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, εσείς τα λέτε θαραλέα, που έχουν αυξήσει τη φτώχεια, που έχουν αυξήσει την ανεργία, που έχουν κόψει κάθε αναπτυξιακή προοπτική, που έχουν κόψει κάθε ελπίδα να βγει η Ελλάδα από την κρίση. Μια, τέτοια προοπτική περιμένει και τις άλλες χώρες που ενδεχομένως εφαρμόσουν τέτοια μέτρα κάτω από τέτοιες πιέσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπερέ, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Προεδρεύον του Συμβουλίου, κύριε Πίτροπε, είναι σύνηθε να χρειάζονται δύο ευρωπαϊκά συμβούλια για να επιλύσουν το θέμα τη ελληνική των κρατών μελών τη Ευρωζώνης προ την Ελλάδα. Ακούω τον κύριο Λάγκερ να ερμηνεύει τη συνθήκη. Ναι, υπάρχει και το γράμμα της συνθήκης, υπάρχει όμως και το πνεύμα. Αν δούμε τα άρθρα 143 και, 180, και 122, οι συντάκτες της συνθήκης δεν είχαν σκεφτεί, κανένας δεν είχαν σκεφτεί ότι πέραν του περάσματος του ευρώ θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα όπως αυτό που έχουμε μπροστά μας σήμερα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε δημιουργικοί και να δείξουμε αλληλεγγύη. Η ιδέα να στείλουμε την Ελλάδα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο φαίνεται για μας που θεωρούμε, που ελπίζουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι και συνεπείς Ευρωπαίοι, τελείως αντίστροφοι λογικά. Κάτι πρέπει να κάνουμε και κάτι πρέπει να ελπίζουμε ως μήνυμα προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι ένα μήνυμα αλληλεγγύης προς την Ελλάδα, ένα μήνυμα ευθύνης σε ό,τι αφορά την οικονομική διακυβέρνηση. Το θέμα αυτό έχει τεθεί επιτάπητος, είναι σοβαρό, είναι ανοιχτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με γαλήνη, να μειώσουμε τις πιέσεις και να ξεκινήσουμε με το ε, και να μην ξεκινούμε με δεδομένο ότι θα πρέπει εξ αρχή να ενισχύουμε ένα εργαλείο που δεν ήταν αποτελεσματικό, το σύμφωνο σταθερότητα, που ήταν κυρίω κατασταλτικό και όχι συνεργατικό. Πρέπει να επιδιώκουμε στόχου για δημόσια ελλείμματα, για χρέη. Χρειαζόμαστε ταυτόχρονα ωστόσο να δημιουργήσουμε πλαίσιο συνεργασία και σωστή προστιθέμενη αξία μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Αυτό, είναι αυτό το ζήτημα είναι στα χέρια των μελών του Συμβουλίου αύριο και ελπίζω να το αντιμετωπίσουν με αίσθημα ευθύνη. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κ. ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τώρα το Συμβούλιο του που έχει χαράξει μια οικονομική, νέα οικονομική στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, εμεί θα πρέπει να αντλήσουμε κάποια συμπράσματα για το φιάσκο τη ε, στρατηγική τη Λισαβόνα. Για να είμαστε ανταγωνιστικοί στι διεθνεί αγορέ, θα πρέπει να είμαστε και καινοτόμοι. Όμω, πολλέ χώρε θα υφίσταν το δυσμενή διάκριση κατά αυτόν τον τρόπο, όπω και η Πολωνία, αλλά και άλλε χώρε τη Ανατολική Ευρώπη, όσο του παροχετευτούν τα κατάλληλα κεφάλαια προ τα εκεί. Στο παρελθόν η Ισπανία, η Πορτογαλία αλλά και άλλε χώρε έχουν ωφεληθεί και έχουν τύχει βοήθειε ε, για τις υποδομές, ε, σιδηρόδρομους, δρόμους, χτίσαν και αυτόν τον τρόπο και αυτό θέλουμε και εμείς να το κάνουμε. Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, πιο συγκεκριμένα έχουμε την, ε, τα, ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το, το, το, Λούμπλιν ας πούμε, θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερες προσοχές στα πλαίσια στρατηγικής για το 2020. Και δεν νομίζω ότι θα ήταν σωστό για αυτές οι φτωχές προχές ε, της Ένωσης να κάθονται και να χρηματοδοτούν την ε, καινοτομία. Ο κύριος Τούσας τώρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρώπη 2020 που συζητιέται σε Σύνοδο κορυφή συνέχεια της στρατηγικής της Λισαβόνας αποδεικνύει ότι τα αντιλαϊκά μέτρα φωτιά που προωθεί η κυβέρνηση του Πασόκ στη χώρα μας με την ουσιαστική συμφωνία όλων των πολιτικών δυνάμεων του κεφαλαίου και των κομμάτων του ευρωμονόδρομου δεν αποτελούν ελληνική ιδιαιτερότητα. είναι προαποφασισμένα από τα πολιτικά επιτελεία και τι κυβερνήσει των κρατών μελών τη ευρωπαϊκή ένωση εντάσσονται στο συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό του κεφαλαίου και προωθούνται με ενιαίο τρόπο σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ένωση με ένταση τη ιδεολογική τρομοκρατία για τη χειραγώγηση του εργατικού λαϊκού κινήματο χρεοκοπούν τα ψέματα οι δημαγωγικέ δηλώσει των εκπροσώπων των αστικών κυβερνήσεων των δυνάμεων του ευρωμονόδρομου ότι η ευρωπαϊκή ένωση η ονε θα αποτελέσουν ασπίδα κατά των κρίσεων τα παραμύθια για την ευρωπαϊκή αγορά των 480 εκατομμυρίων τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια την κοινοτική αλληλεγγύη και άλλα τέτοια ιδεολογήματα η ευρωπαϊκή ένωση είναι η υπεραλιστική διακρατική ένωση του κεφαλαίου των μονοπωλίων που με ενιαία στρατηγική επιτίθενται στους λαούς και διασταυρώνουν τα μαχαίρια τους για τη μοιρασιά της λίας. τα οικονομικά πολιτικά προβλήματα στην ελλάδα στα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης θα λυθούν με την πάλη του εργατικού λαϊκού κινήματος την πάλη και την αλληλεγγύη των λαών. είναι προφανές ότι αυτό που γίνεται στην ελλάδα έχει να κάνει σχέση με τον έντονο διαγωνισμό που γίνεται μεταξύ των υπεριαλιστικών κρατών και μεταξύ της ευρωπαϊκής ένωσης των ηπα της κίνας και άλλων αναπτυσσόμενων χωρών. έτσι μπροστά και απέναντι στη στρατηγική του κεφαλαίου η εργατική τάξη τα λαϊκά στρώματα επιβάλλεται να αντιτάξουν τη δική του στρατηγική πάλι για την ανατροπή αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής προκειμένου να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Ευχαριστώ. Ο κύριο Χόκμαρ για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Δύο τι να θέλω να σα αναφέρω κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά και δεύτερον για την ανταγωνιστικότητα. Πέρσι τέτοια εποχή συζητούσαμε εδώ στο Κοινοβούλιο πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Και κάποιοι έλεγαν μεγαλύτερες δαπάνες ε, παρά τα μεγάλα ελλείμματα. Άλλοι, εμείς λέγαμε σταθερότητα δημόσιες δαπάνε και συγκράτηση του ελλείμματο. Να τα αποτελέσματα τώρα κάποια κράτη-μέλη ακολούθησαν αυτή την πολιτική των δαπανών και την αποδοχή των μεγαλύτερων ελλείμματων και του γινόμαστε μάρτυρες των συνοποιών. Αύξηση του δημοσίου χρέου, αύξηση των δαπανών εξυπηρέτηση για την μια που αυξήθηκαν τα επιτόκια να πάνε στις εξυπηρέτησης του χρέους. Να τι θα πρέπει να, να προσέξουμε, να μην κάνουμε τα ίδια λάθη με τα περισσότερα κάτι μέλη και άρα θα πρέπει να αντιλήσουμε κάποια μαθήματα από τη συγκυρία ότι δηλαδή θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες που ήδη ισχύουν και επίσης θα πρέπει να δούμε πώς το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης θα θωρακιστεί, θα περιχαρακωθεί για να αντιμετωπίσει και τις μέλουσες κρίσεις. Μερικοί λένε τώρα θα πρέπει τη στατική εξόδου να την ε, αναβάλουμε, να την καθυστερήσουμε και σε σχέση με την καθυστέρηση εξυπηρέτηση του ελλείμματο. Ε, αυτό είναι λάθο, γιατί αυτό μα υπονομεύει την δυνατότητα τη ε, ανάκαμψης και αυτό πρόκειται να εκτινάξει ακόμη περισσότερο τα επιτόκια. Η ιδεα ε, ανταγωνιστικότητα πάει χέρι-χέρι με τη δυνατότητα των σταθερών δημοσίων οικονομικών και τη δυνατότητα του να επιφέρουμε τις πραγματικές ε, αλλαγές που χρειάζονται εδώ και δεκαετίε. Να, επομένω ποια είναι η πρόκληση για το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούλμαν, δύο λεπτά έχει το λόγο. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, αξιότιμοι συνάδελφοι Χουεκμάρκ. Πιστεύω ότι τις τελευταία χρόνια στα... ήμασταν σε άλλα κοινοβούλια. Γιατί εγώ άλλο κοινοβούλιο γνώρισα από αυτό που περιγράφεται. Έζησα το κοινοβούλιο όπου είπαν ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε ε, ε, τα hedge funds, τα ιδρύματα αξιολόγησης επιστολεπτικής ικανότητας θα πρέπει να κοιτάξουμε τα κρίσιμα προϊόντα, τους κρίσιμους οικονομικούς φορείς προκειμένου να μην καταλήξουμε σε διεθνές φιάσκο και άλλοι μας έλεγαν ότι μα αφήστε τα αυτά και μην ασχολείστε, τα ρυθμίζει από μόνη της η αγορά και ο κύριος Μαγκρίβη τελικά είδαμε ποιο είναι το αποτέλεσμα είδαμε το διεθνές φιάσκο που ευθύνεται για την υπερχρέωση των κρατών μελών και είναι πραγματικά απίστευτο ότι σήμερα ερχόμαστε και λέμε ότι είναι λάθος η κατεύθυνση της πολιτικής απασχόλησης. Μιλάμε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση με, τα, με τη συζήτηση αυτή και εδώ που μας λέει ο συνάδελφος Λάγκεν ότι η κυρία Μέρκελ ε, κατάλαβε τις ευρωπαϊκές συνθήκες, όχι μόνο που την κατάλαβε την ευρωπαϊκή συνθήκη, αλλά ακόμα χειρότερα είναι σε θέση να υπονομεύσει τις ευρωπαϊκές συνθήκες και αυτά που συνεπάγονται για να μην χάσει ε, μια σημαντική ψηφοφορία. Αλλά αυτή δεν είναι η αντιμετώπιση που χρειαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπαμε ότι είναι πολύ αποδυναμωμένη η στρατηγική το 2020 να μας αποδείξετε ότι μπορείτε να κινητοποιήσετε νέα μέσα, να καταπολεμήσετε, για, να πολεμήσετε μάλλον για πιο πολλές δυνατότητες ανάπτυξης στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουν μια ευκαιρία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ας ε, δημιουργήσουμε λοιπόν ευρωπαϊκά μέσα αυτό αποτελεί το βασικό μας μήνυμα προς την Σύνοδο, γιατί μόνο τότε μπορεί να ελπίζει ο κόσμος ότι θα δώσουμε τις σωστές απαντήσεις. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Βέιμπερ για ένα μισή λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, ο συνάδελφος Σούλτς μας παρουσίασε ότι η Ελλάδα ε, έχει παραδοθεί στα νύχια. Δηλαδή, τι, η Ευρώπη πρέπει να λέει και ευχαριστώ αν κάποια κράτη-μέλη δεν έχουν τηρήσει τους κανόνες του παιχνιδιού και πέρσι που έλαβε μέτρα σκληρά η Ιρλανδία κανείς δεν ε, είπε ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Κυρίες και κύριοι, φυσικά αντιμετωπίζουμε μεγάλη πίεση, αλλά το γεγονός είναι ότι η Ελλάδα αντιμετώπισε τεράστια ε, προτερήματα, ωφέλησε ό,τι αφορά τα επιτόκια κατά την εισχώρηση στην Ευρωζώνη. Τα έφαγε όμως η Ελλάδα αυτά τα πλεονεκτήματα. Ποιος είναι ο καλός Ευρωπαίος, αυτός που βάζει λεφτά και δίνει λεφτά στο τραπέζι σήμερα. Όχι, αυτός ο οποίος εφαρμόζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Αυτός είναι ο καλός Ευρωπαίος. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ενισχύσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί οι προτάσεις ε, οι μακροπρόθεσμες που έχει υποβάλει κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε μία ε, ισχυρή επιτροπή που θα ελέγχει το 3%, το κανόνα του 3% γιατί δεν καταφέραμε στην Ευρωζώνη να τηρήσουμε το 3% και να σκίσουμε και το σχετικό έλεγχο. Άρα ναι, υπέρ μια ισχυρού επιτροπή που θα μπορέσει να το τηρήσει αυτό στο μέλλον. Για να μιλάμε θετικά και για το ευρώ. Γιατί δεν είναι κρίση νομίσματος, είναι οικονομική η κρίση που αντιμετωπίζουμε. Και τελικά θα πρέπει να ωφεληθεί το ευρώ. Άρα ναι για το ισχυρό αυτό νόμισμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λέινεν, 1,5 λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κρίση στην Ελλάδα είναι ένα επίκαιρο πρόβλημα, αλλά η κρίση στο περιβάλλον είναι μακροπρόθεσμο πρόβλημα και τα δύο θα πρέπει να επιληθούν με την επίλυση μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στη στρατηγική του 2020 αναφέρθηκε ότι θα πρέπει η ανάπτυξη να είναι βιώσιμη και ενοποιημένη. Κοιτώντα όμω τι συστάσει του Συμβουλίου, τα πράγματα είναι πολύ πιο περιορισμένα. Περιορίζονται στι κλασικέ ε, ε, στρατηγικέ ανάπτυξη, οι οποίε απέτυχαν. Δεν μπορεί να είναι ευφυή η ανάπτυξη αν δεν είναι βιώσιμα και δεν μπορεί να είναι ευφυής αν δεν είναι ενοποιημένη. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ από την Προεδρία να φροντίσει αυτό το τρίπτυχο, αυτοί οι τρεις πυλώνες να παραμείνουν, γιατί αυτό είναι το καινοτομό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Είμαι πολύ ευχαριστημένος ε, για το γεγονός ότι οι πόροι, ότι προωθείται μάλλον ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ανάπτυξη με την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας για να μειώσουμε την εξάρτηση, να μειώσουμε το κόστος, να λύσουμε μια σειρά προβλημάτων. Αναμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας υποβάλει το 2010 ένα σχετικό οδικό χάρτη, γιατί είναι μεικτή αυτή η εργασία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μέλων και πολλά ακόμα είναι ασαφή. Θα πρέπει λοιπόν να οριστούν συγκεκριμένες μευτικοί στόχοι, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον στόχο της ε, εξοικονόμησης, του 20% της ενέργειας προκειμένου να κάνει και η βιομηχανία τις σχετικές επενδύσεις που χρειάζεται. Ο κύριος Μάουρο, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν μου θέτατε την ερώτηση που κάνουν συχνά στην Ιστινία θα έλεγα θα έλεγα σε τι χρησιμεύει η Ευρώπη και η απάντηση θα έρχονταν από το βάθος καρδίας μου. Μόνο για να βοηθήσει την Ελλάδα κάτω από τις παρούσες συνθήκε. Δεν είναι παραλογισμός να το σκεφτούμε. Στο DNA, στη φύση του ευρωπαϊκού πολιτικού εγχειρήματο υπάρχει η αλληλεγγύη. Με πλήττει ταυτόχρονα ωστόσο το γεγονός ότι αυτοί που λένε ότι θέλουν να χτυπήσουν την οικονομική κερδοσκοπία θέλουν να την υποκαταστήσουν με την πολιτική κερδοσκοπία. Πώς μπορεί κανείς να σκεφτεί, για παράδειγμα, να ε, διεξάγει τη μάχη αυτή κόντρα στην καγκελάριο Μέλκελ. Να σκεφτεί δηλαδή ότι ο στόχος της προσπάθειας υποστήριξης με αλληλεγγύη της Ελλάδος σημαίνει να υπάρξει επίθεση σε ένα άλλο κράτος μέλος. Γιατί μας θυμίζει με απλά λόγια ότι η πολιτική αλληλεγγύης πρέπει να συνοδεύεται και από μια πολιτική ευθύνη. Είναι ένα αίτημα που πολλές φορές το κάναμε. Γιατί ξέρουμε ότι μέσω αλληλεγγύης και ευθύνης θα πετύχουμε να καταστήσουμε ε, λογικό και ε, να αγγίξουμε όλους με, για το ευρωπαϊκό πολιτικό εγχείρημα. Ότι στόχος μας είναι κυρίως να προωθήσουμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας, μας, μας χωρίζουν. Πρέπει λοιπόν η Ένωση να είναι φιλόδοξη και να απαιτήσει από τα κράτη-μέλη την ε, αυστηρότητα που θα απαιτηθεί για να μπορέσει μακροπρόθεσμα να υλοποιηθεί με αλληλεγγύη και με ευθύνη το ευρωπαϊκό πολιτικό σχέδιό μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κοφεράτη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ελληνική κρίση είναι αντικειμενικά το σοβαρότερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Και προκύπτει προφανώς από την έλλειψη ορθού τρόπου διαχείρισης των δημοσίων δαπανών. Είναι ακατανόητη τόσο η καθυστέρηση με την οποία παρεμβαίνουν τα ευρωπαϊκά όργανα για να ενισχύσουν ένα κράτος μέλος αυτή τη στιγμή δυσκολίες. Και η καθυστέρηση αυτή είχε ήδη αρνητικέ συνέπειες. Άφησε αντικειμενικά χώρο στη δράση των κερδοσκόπων. Δημιούργησε στο εσωτερικό της Ένωσης αμφιβολίες για την αλληλεγγύη κάποιων χωρών σε ό,τι αφορά το μέλλον της Ευρώπης. Μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για το πρώτο μεγάλο πρόβλημα που καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε μετά την θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Επιδίνωσε τις δυσκολίες της ελληνικής κυβέρνησης που χρειάστηκε να υιοθετήσει μη δημοφιλή μέτρα που δεν προκύπτουν που έχουν σημαντικές συνέπειες για εκατομμύρια πολιτών χωρίς να είναι βέβαιοι ότι θα ερχόταν η βοήθεια. Επιπλέον, αντικειμενικά έθεσε σε κίνδυνο την βασική αρχή της ελεγγύης που ήταν μια, ένα κοινό μέλλον για όλη την Ευρώπη. Είναι αναγκαίο λοιπόν να υπάρξει παρέμβαση χωρίς καμία κερδοσκοπία. Να θυμίσω στον κύριο Μάουρο ότι η Γερμανία είναι αναμφίβολα μεταξύ των χωρών που, είχαν, που έχουν κερδίσει περισσότερο από την θέση σε ισχύ του ευρώ και από τι σχέσει που δημιουργήθηκαν με τα επιτόκια. Πρέπει να αναλάβουμε δράση γρήγορα για να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Αυτό πρέπει να το κάνει η Ευρώπη προ το συμφέρον τη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ο κύριο Μαρινέσκου για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το Συμβούλιο με ενθουσιασμό δέχτηκε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη στρατηγική για το 2020. Γιατί χρειαζόταν ένα τέτοιο έγγραφο και γι' αυτό θα αξίζει πάρα πολύ μεγάλης προσοχής και όσον αφορά την οικονομική αρρωγή θα πρέπει να συνοηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τα κονδύλια ε, και την ε, πιο δόκιμη χρήση τους. Κατά τη γνώμη μου δεν θα πρέπει να κάνουμε τίποτα με τον προϋπολογισμό πριν ε, προσέξουμε την ΚΑΠ αλλά και την πολιτική της συνοχής. Ανάπτυξη, σταθερότητα χρειάζεται και επομένως χρειάζεται έργα υποδομής στην ενέργεια και στις μεταφορές. Δεν έχει προσεχτεί αυτό στο έγγραφο το τι θα γίνει σε αυτούς τους τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα εναρμονίσουμε την υποδομή μας με τις ε, χώρες. Αυτό πρόκειται να μας οδηγήσει σε μια ανάπτυξη βιώσιμη, θα μας οδηγήσει σε θέσεις απασχόλησης και έτσι θα καταφέρουμε την, την ασφάλεια που χρειάζεται όσον αφορά την προμήθεια της ενέργειας αλλά και την ασφάλεια στις μεταφορές. Γι' αυτό και θα πρέπει να ζητήσουμε από το Συμβούλιο, να ζητήσει από την Κομισιόν να κατεβάσει κάποιες προτάσεις σε αυτό το τόσο σημαντικό τομέα για την στρατηγική του 2020 και αυτό θα είναι προς το συμφέρον όλων των Ευρωπαίων. Ε, Η κυρία Ποδηματά για δύο λεπτά. ευρωπαϊκού συμβουλίου τη 11 η φεβρουαρίου που ήταν να στείλει ένα μήνυμα υποστήριξη στην ελλάδα ώστε να ηρεμήσουν οι αγορές έχει στην ουσία ακυρωθεί εξαιτία τη κακοφωνία και τη αβεβαιότητας που επικράτησε στου κόλπους της ευρωπαϊκής ένωσης. το ευρωπαϊκό συμβούλιο που αρχίζει αύριο τις εργασίες του δεν έχει καμία πολυτέλεια να διατηρήσει το σημερινό κλίμα αβεβαιότητας και κακοφωνίας οι πάντες αναγνωρίζουν πλέον ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρει πολύ σκληρά μέτρα τα περισσότερα από τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται με κόστος και θυσίες από τον ελληνικό λαό. όμως την ίδια ώρα συνεχίζει να δανείζεται με εξαιρετικά υψηλά επιτόκια με τελευταίο παράδειγμα αυτό της 5ης μαρτίου γιατί υπάρχουν κερδοσκόποι στις αγορές που κάνουν περιουσίες στοιχηματίζοντας τις πιθανότητες χρεοκοπίας μιας χώρας και εν τέλει δημιουργώντας τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό. σήμερα η συζήτηση αφορά στην ελλάδα αύριο ενδεχομένως να αφορά σε ένα άλλο κράτος μέλος. θα το σταματήσει αυτό το ευρωπαϊκό συμβούλιο δημιουργώντας έναν ευρωπαϊκό αποτελεσματικό αποτρεπτικό μηχανισμό που θα θωρακίσει τις εθνικές οικονομίες και τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ. μίλησε ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής επιτροπής για ευθύνη και αλληλεγγύη και είχε δίκιο χρειάζονται και τα δύο όταν συμμετέχει κανείς σε μια οικογένεια όπως είναι η ζώνη του ευρώ. αλλά δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που να αμφιβάλλει ότι η ελλάδα έχει πλήρως αναλάβει τις ευθύνες της αλλά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της σε αυτή τη δύσκολη φάση τα θηρία των αγορών. πριν από ενάμιση χρόνο οι αγορές απείλησαν με κατάρρευση την παγκόσμια οικονομία. δεν θα απειληθεί η ελλάδα σήμερα; εδώ λοιπόν έρχεται η έννοια της αλληλεγγύης που θα έπρεπε να είναι αυτονόητη και σύμφυτη με τη συμμετοχή στο ευρώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σβάμπ, για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, για την Ελλάδα ακούσαμε ήδη πάρα πολλά. Θα ήθελα να στρέψω το βλέμμα μου στο μέλλον και να δούμε τι θα γίνει με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έθεσε ένα σημαντικό έγγραφο που θα αποτελέσει και τις κατευθυντήριες γραμμές για τις βασικές πολιτικές της Ένωσης. Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι οι κοινοί στόχοι τους οποίους ορίσαμε στην ε, στρατηγική το 2020 θα πρέπει να τους ακολουθήσουμε. Αυτό αποτέλεσε μεγάλο πρόβλημα στη συνθήκη της Λισαβόνας, στη στρατηγική της Λισαβόνας. Και θα πρέπει να το επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό. Μόνο αν τηρήσουν όλα τα κράτη-μέλη τους ορισμένους στόχους, θα μπορέσουμε πραγματικά να τους πετύχουμε αυτούς τους στόχους από κοινού. Και αυτό δεν θα το πετύχουμε αν ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, αντιλαμβάνεται το ρόλο του ως διοικητικό ε, μόνο όργανο για την, τελευταία στιγμή, την εφαρμογή τελευταία στιγμή των κανόνων. Και συνάδελφοι θα το πετύχουμε αυτό μόνο αν η αρχή της αλληλογγύης ορίζεται βασικά σε αυτή τη στρατηγική του 2020. Αυτό τι σημαίνει η ίδια ευθύνη των κρατών μελών για όλους τους τομείς όπου πραγματικά έχουν ευθύνη και σε αυτό συγκαταλέγεται και ο δημοσιονομικός απολογισμός, αλλά φυσικά θα πρέπει να υπάρχει και υποχρέωση συνδρομής για τα άλλα κράτη-μέλη σε περίπτωση ανάγκης και αυτό, συνάδελφοι, θα το πετύχουμε μόνο αν η πολιτική ηγεσία ασκηθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία τα σφάλματα που κάναμε στη στρατηγική της Λισαβόνας. Γιατί ακούσαμε πολλές φορές ότι η στρατηγική της συνεργασίας απέτυχε σε ό,τι αφορά τη στρατηγική της Λισαβόνας. Χρειαζόμαστε λοιπόν σαφείς στόχους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία θα στηρίξει, την οποία θα στηρίξει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, ε, Ο κύριος Πουπάκης θέλει το λόγο. Με, μπλου, με μπλε κάρτα. Όχι. Όχι. Με συγχωρείτε. Ο κύριος Λόπες Αγγιγιάρ έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι έχουμε επίγνωση του ότι 500 εκατομμύρια πολιτών παρακολουθούν με ασυνήθιστη προσοχή τα, το τι θα γίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Διότι θα μπορέσει να δώσει ένα μήνυμα εξόδου από την κρίση που είναι αυτό που περιμένουν οι πολίτες ε, Κυρίω, η έξοδος από την, θα, την κρίση θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται μέσα στη στρατηγική του 2020. Μια πλήρη προσέγγιση ανάπτυξης κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής. Από την οπτική γωνία της διακυβέρνησης και από την οπτική γωνία της προστασίας των εργαζομένων, της κοινωνικής προστασίας και της διαφύλαξης του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και της ισότητας. Και θέλω να τονίσω ένα κείμενο που μπορεί να βελτιώσουμε την έννοια της ε, ισότητας. Την, ε, τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη έγινε, πήρε την ηγετική θέση στην προστασία της, ε, του κλίματος και την μάχη για την μείωση των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος με την, και που θα μειώσει την απογοήτευση με την οποία φύγαμε από την Κοπενχάγη. Βάση όλων πιστεύω είναι ότι στο Συμβούλιο πρέπει να υπάρξει μια σαφής ευρωπαϊκή απάντηση για, την, για να συνοδεύσει την ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική με δημοσιονομικές και φορολογικές προσεγγίσεις στο ύψος της Ευρώπης. Το μήνυμα της ελληνικής για την Ελλάδα δεν είναι ένα μήνυμα για την Ελλάδα, είναι ένα μήνυμα για την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους. Δεν θα διασώσουμε την Ελλάδα. Θα δώσουμε μήνυμα ευρωπαϊκής ζωής για την βασική αυτή πρόκληση, για τη βασική αυτή επιλογή που κάναμε με την ΟΝΕ. Και δεν μιλάμε για την Ευρώπη, μιλάμε για όλους. Υπήρξε καθυστέρηση απάντησης από τα θεσμικά όργανα. Δεν πρέπει να υπάρχει καθυστέρηση στην απάντηση, στην υλοποίηση των αποφάσεων του επερχόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ξεκινούμε τη διαδικασία Catch the Eye. Το λόγο έχει για ένα λεπτό κάθε αγωδητής. Ξεκινάμε με τον κύριο Κάστερ. Αν δεν είναι εδώ ο κύριος Κάστλερ, το λόγο έχει Το λόγο έχει ο κύριος Λούαν. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Κουμουτσάκος. Πού είναι εδώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι αλήθεια ότι η χώρα μου η Ελλάδα διαχρονικά δεν ανέπτυξε όταν και όσο έπρεπε την οικονομία της. Με μέτρο και με σύνεση Τώρα έχει αναλάβει όμω πλήρω τι ευθύνε τη. Ο ελληνικό λαό καταβάλει δυσβάστακτο τίμημα. Α μην κρυβόμαστε όμω. Η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα τη ΩΝΕ που αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Δεν ήταν η μόνη που προσέφυγε στι δηλητηριώδει υπηρεσίε γνωστών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Δεν είναι ούτε θα μείνει ο μόνο στόχο των κερδοσκόπων. Όλοι γνωρίζουμε και το γνωρίζουμε καλά ότι το ελληνικό ζήτημα είναι και ευρωπαϊκό ζήτημα. Η ΟΝΕ θα μείνει ακροτηριασμένη χωρί περισσότερο συντονισμό οικονομική και φορολογική πολιτική και πάνω απ' όλα χωρί αλληλεγγύη. Η κρίση, κάθε κρίση είναι μητέρα αλλαγών. Η σημερινή κρίση μπορεί να γεννήσει μια ισχυρότερη Ευρώπη και η Ελλάδα μπορεί να είναι η μέα αυτή τη αλλαγή. Α μην πυροβολούμε λοιπόν την Ελλάδα. Α πυροβολήσουμε όλοι μαζί του κερδοσκόπου που θα ήθελαν να δουν ένα γονατισμένο ευρώ. Και αυτό οφείλει να πράξει το αυριανό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Σταμπάτζη έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να επιστήσω την προσοχή του Συμβουλίου και τη Επιτροπή ότι υπάρχουν μια σειρά για την πολιτική και στατική του 2020 αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι ισχύουν τώρα εύρυθμα λειτουργούσε πολιτικέ όπω η ερωτική πολιτική. Οπότε με κάποια μεταρρύθμιση είναι δυνατόν να μας βοηθήσουν αυτές οι πολιτικές να πετύχουμε τους στόχους με το 2020. Επίσης θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο τις πολιτικές μας που ήδη λειτουργούν καλά. Και αν θέλουμε στην ιστορία να έχουμε εναρμόνιση, θα πρέπει να σκεφτούμε την, τις υποδομές, την ενέργεια, την ασφάλεια των προμηθειών, περισσότερους πόρους να κατευθύνουμε προς ε, αυτές τις πολιτικές. Περισσότερες μεγαλύτερες δαπάνες. Όλα θα πρέπει να συζητηθούν σωστά και επομένω θα πρέπει να προσέξουμε την πολιτική της συνοχής και να λάβουμε υπόψη και τις περιφέρειες της Ευρώπης. Και τώρα. Ο κύριος το Τόιρερ, για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση για το ευρώ, η συζήτηση για την Ελλάδα ε, τις τελευταίες ημέρες ε, επικράτησε ιδιαίτερα και κυριέρχησε. Με ανησυχεί το γεγονός ότι στη Γερμανία σήμερα 40% των Γερμανών λένε ότι η εισαγωγή του ευρώ ήταν σφάλμα. Αυτό θα πρέπει να μας ανησυχεί, γιατί δεν είναι μονόδρομο στο κοινό νόμισμα, δεν πρόκειται για μια ανεπιστρεπτή διαδικασία και θεωρώ ότι η υπόσχεση που δώσαμε σε ό,τι αφορά το ευρώ, ότι θα πρέπει να είναι δηλαδή εξίσου δυνατό όπως το Μάρκο, θα πρέπει να την τηρήσουμε και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι στην Ευρώπη χρειαζόμαστε μια συζήτηση για την κοινωνική ε, οικονομία της αγοράς. Δεν θα πρέπει να συζητήσουμε πώς μπορούμε να κάνουμε τη Γερμανία λιγότερο ανταγωνιστική. Θα πρέπει να συζητήσουμε πώς όλη η Ευρώπη θα πρέπει να καταστεί ανταγωνιστική προκειμένου να σημειώσει επιτυχία και στις παγκόσμιες αγορές. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ μια συζήτηση τέτοια για την κοινωνική οικονομία της αγοράς στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λούνατσεκ, η κυρία Λούνατσεκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με εκείνους που ζητούν μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση σε ό,τι αφορά τον οικονομικό τομέα, ιδιαίτερα σήμερα. Ελπίζω αυτό να συζητηθεί όχι μόνο στη Σύνοδο για την Ευρωζώνη, αλλά και στο ιστορικό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ωστόσο, και το είπε ο συνάδελφο πριν από λίγο, υπάρχει και ο αρνητικό αντίκτυπο, ο οποίο διατυπώνεται από τον κόσμο. Υπάρχει ένα εγγενέ λάθο και σφάλμα στην Ευρωζώνη με στο κοινό νόμισμα. Πώς μπορούμε να έχουμε κοινό νόμισμα χωρίς να έχουμε κοινή οικονομική πολιτική. Αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος. Θα πρέπει να ακούσουμε τη φωνή τη λογική και η δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Αυτό επιτάσσει η φωνή της λογικής για την υποστήριξη της Ελλάδας. Αλλά αυτό που λέω και δεν ακούω στη συζήτηση είναι ότι και η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει πολλά για παράδειγμα, να περικόψει τις στρατιωτικές δαπάνες. Μία ευρωπαϊκή χώρα η οποία δίνει άνω το 4% σε τέτοιες στρατιωτικές επενδύσεις από τη Γερμανία, από τη Γαλλία, όλα αυτά τα χρειαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί θα πρέπει να γίνουν επίσης περικοπές. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μπάφτον. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα διορθώσουμε αυτά το βράδυ στο πρωί. Όλοι εδώ ανέφεραν το πρόβλημα τη Ελλάδο και έρχεται ο κ. Μπαρόσο και μα λέει ότι για αυτό το διήμερο συμβούλιο το θέμα δεν είναι καν στη μερισσία διάταξη. Είναι απίστευτο αυτό, μια που όλο ο κόσμο ε, να ταινίζει προ τα εδώ να δει τι θα αποφασίσουμε και βλέπουμε ότι θέλουμε απλώς να τα κουκουλώσουμε, να κουκουλώσουμε το ότι η Ευρώπη δεν τα πάει καλά και ότι έχει πάρει την κατηφόρα. Α, οι Γερμανοί τι λένε, είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι. Όμως δεν θα πρέπει να καπελώνουμε τους Έλληνες, θα πρέπει αυτοί να αποφασίζουν, ίσως να κάνουν ένα δημοψήφισμα αν θέλουν να έχουν το ευρώ. Είναι δική τους υπόθεση και με αειδιάζουν αυτές οι εγωιστικές απόψεις των κρατών που φροντίζουν μόνο του οίκου τους. Και η Ισπανία και η Πορτογαλία και η Ελλάδα για όλους το ίδιο ισχύει. Θυμηθείτε τα λόγια μου. Το πρόβλημα το σημερινό θα υπάρξει για αύριο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπρόνς, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα προβλήματα της Ελλάδας και της Ευρωζώνης δεν πρέπει να θεωρηθούν ω εξαίρεση. Ένα ενιαίο νόμισμα για, ένα τόσο μεγάλο ετερογενή, για μια τόσο μεγάλη ετερογενή περιοχή της Ευρώπης είναι προβληματικό. Η αξία ενός νομίσματος αντικατοπτρίζει την οικονομία της περιοχής. Όταν πάει καλά η οικονομία, η αξία του νομίσματος ανεβαίνει. Όταν η οικονομία ε, πέφτει σε ύφεση, το νόμισμα ε, υποτιμάται. Η κατάσταση της Ελλάδος ε, οδήγησε σε μείωση, θα οδηγούσε σε μείωση, σε υποτίμηση του νομίσματος της, κάτι που θα ήταν θετικό γιατί θα μπορούσε να έχει αύξηση του τουριστών. Η Ευρώπη δεν είναι η λύση στα οικονομικά προβλήματα του κόσμου, αλλά το πρόβλημα. Η δυσκολία της Ελλάδας είναι ότι αν έφευγε από το ευρώ τώρα θα αντιμετώπιζε ε, πολλαπλασιασμό του χρέους της ε, ε, στο ευρώ και θα ήταν μια απειλή για την ευρωζώνη. Αυτό θα πρέπει να ε, είναι μια προειδοποίηση για τι χώρε που δεν είναι στο ευρώ. Προσοχή, έτσι και μπείτε μέσα, είστε κλειδωμένοι εκεί για πάντα. Ευχαριστώ. Η κυρία Φλασίκοβα για ένα λεπτό. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπρόεδρε, θα είμαι σύντομη. Τα περισσότερα έχουν ήδη υποθεί. Άποψή μου είναι ότι η κατάσταση που συζητούμε τους τελευταίους μήνες, η Ελλάδα δηλαδή, δεν είναι μοναδική η κατάσταση. Από ό,τι φαίνεται, η ιδέα προχωρούμε προ την ιδέα μια νέα αντιμετώπιση του Συμφώνου σταθερότητα και ανάπτυξη. Είτε θα παραμείνουμε στην τήρηση του γράμματο των συνθήκων, είτε θα δεχθούμε ότι το Σύμφωνο σταθερότητα πρέπει να προσαρμοστεί. Και σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να γίνουν οι προσαρμογές με τέτοιο τρόπο που θα μας επιτρέψουν να διαφυλάξουμε την οικονομική σταθερότητα και την ανάπτυξη όχι μόνο στις χώρες της Ευρωζώνης αλλά που σε τρόπο που θα επιτρέπει και σε χώρες εκτός της Ευρωζώνης να ενταχθούν στην ζώνη του ευρώ χωρίς να χρησιμοποιούνται ε, στις χώρες αυτές πόροι διαδοτικών ταμείων. Ευχαριστώ. Grazie. La parola all'onorevole per un minuto. Ο κύριο Οντί, για ένα λεπτό. Μία παρατήρηση και τρεις προτάσεις, πρόεδρε. Πρώτον, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έρχεται ο κύριος Βαν σε μία σύνοδο τόσο σημαντική. Ε, θα έπρεπε να είναι παρόν. Τρει προτάσει για την ανάκαμψη της Ευρώπης. Μέσω πρόθεσμα υποστηρίζω την ιδέα του κύριου Κονμπέντιτ που, έγινε, που την υιοθέτησαν και άλλοι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούσε να κάνει ένα σύμφωνο με την Τουρκία για την επίλυση του Κυπριακού, θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε κατά 2% το ΑΕΠ της Ελλάδος. Άλλη οικονομική πρόταση, δεν έχουμε τα εργαλεία αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν ε, εγγυάται η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να δεσμεύσει πόρους τα δάνεια τη Ελλάδα, κάτι που θα μείωνε σημαντικά το κόστο για την Ελλάδα. Τρίτον, λένε ότι ήταν ψεύτικοι οι προπολογισμοί. Δεν συμβαίνει μόνο αυτό στην Ελλάδα αυτό. Α κάνουμε συγκεκριμένου λογιστικού κανόνε για όλα τα κράτη τη Ένωση, ώστε να έχουμε λογαριασμού τακτικού, ειλικρινεί και σωστού για όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Λυπούμε. Έχουμε και άλλα δέκα αιτήματα στο πλαίσιο του Catch the Eye. Θα διακόψουμε ωστόσο για να δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή. Παρακαλώ τον Επίτροπο κ. Σεύκοβιτς να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς να πω πόσο με εντυπωσίασε η σαφή ε, επίδειξη ελληνική και από τις εκκλήσεις για ανάληψη ευθυνών που ακούσαμε από τους πιο πολλούς ομιλητές. Ακριβώς αυτό χρειαζόμαστε στην παρούσα φάση, γιατί είναι σαφές ότι το ευρωπαϊκό πρόβλημα χρήζει ευρωπαϊκής λύσης. Και πολλές φορές αναρωτιέμαι μήπως δεν έχουμε μάθει αρκετά από το παρελθόν και ποιο θα ήταν ο αντίκτυπος αυτό για το μέλλον μας αν δεν ακολουθήσουμε δηλαδή ευρωπαϊκές λύσεις για ευρωπαϊκά προβλήματα αν ε, θέλουμε να βρούμε συλλογικέ λύσει. Είναι σαφέ ότι δεν είμαστε μόνο μία ομάδα χωρών, είμαστε μια ευρωπαϊκή οικογένεια και όταν ε, ένα μέλο τη οικογένεια έχει πρόβλημα θα πρέπει να το βοηθήσουμε. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να προτείνει ένα μέσο συντονισμένη ε, συνδρομή στην Ελλάδα απόλυτα συμβατό με το ευρωπαϊκό δίκαιο και είμαι βέβαιο ότι αυτό είναι δυνατόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την υποστήριξη σε της στρατηγικής για το 2020. Δεν θέλω να επαναλάβω, αλλά θέλω να τονίσω πόσο αναμένουν οι Ευρωπαίοι πολίτες αυτή την ηγεσία, πόσο θέλουν να βελτιώσουμε την απόδοσή μας, πόσο περιμένουν να τους καθοδηγήσουμε μετά την κρίση. Θα θέσουμε λοιπόν πολύ σαφείς μεσοπρόθεσμους στόχους σε ό,τι αφορά και τους εταίρους μας όπως ε, η η, η Κίνα, η Ινδία. Νομίζω ότι έχει έρθει ο χρόνος, η χρονική στιγμή για να λεφθούν αποφάσεις. Άκουσα τις εκκλήσεις για καλύτερη διακυβέρνηση, άκουσα τις εκκλήσεις για καλύτερη οικονομική και χρηματοοικονομική εποπτεία, ότι θα πρέπει να εφαρμόσετε καλύτερα το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αυτό ακριβώς έχει κατά νου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θα αποτελέσει το στόχο των προτάσεων που σύντομα θα ακολουθήσουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας, όλους όσοι υποστήριξαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την υποβολή σαφών στόχων στις ε, συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αύριο. Είναι σημαντικό να υπάρχει μεσοπρόθεσμη στρατηγική θεωρώ, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και σαφείς δείκτες. Σαφείς δείκτες. Προς τα πού κινούμαστε, ποιοι είναι οι στόχοι μας. Και γι' αυτό λοιπόν επιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αποδεχτεί αυτούς τους συγκεκριμένους στόχους μετά τι διαβουλεύσεις της αυριανής και μεθαυριανής ημέρα. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη απασχόληση, καλύτερη διάσταση των δύο φύλων, καλύτερη εκπαίδευση και σαφώς χρειάζεται να επενδύσουμε περισσότερο στην έρευνα και στην ανάπτυξη και σαφώς χρειάζεται να καταπολεμήσουμε την ένδυα. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμένει σε θέματα αλληλεγγύης, ευθύνης, συγκεκριμένης στρατηγικής για την Ευρώπη και για τον Ευρωπαίο πολίτη. Θα ήθελα να εκφράσω στο σημείο αυτό την ελπίδα μου, αυτό το θετικό πνεύμα το οποίο παρουσιάστηκε εδώ υπέρ της αλληλεγγύης και της ανάληψης ευθενών να είναι εξίσου διακριτό και στις διαβουλεύσεις των αρχηγών μας αύριο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε και τώρα. Θα το λόγο για του Συμβουλίου. Ο Υπουργό κ. Λόπεθ Γκαρίδο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέει στα Ιταλικά ο Υπουργό. Ήταν πολύ σημαντική η συζήτηση που έγινε γιατί αφορούσε ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ανησυχίας αυτό η κρίση για την Ελλάδα Γίνεται κάτι που όπως σωστά είπε ο κύριος Σοντή ορθώς έγινε εδώ σε ε, παρουσία του Συμβουλίου μα ε, το Συμβούλιο εγώ εκπροσωπώ και σε σχέση με το πρόβλημα της Ελλάδας το πλήστον συζητήθηκε σήμερα εδώ είναι κάτι για το οποίο έχουμε ξεκάθαρες ιδέες ως Συμβούλιο. Η Ευρώπη αφορά την ολοκλήρωση από πλευράς και οικονομικών πολιτικών. Αλληλεγγύη. Κοινωνικό περιεχόμενο. Δεύτερον. Και κατά τρίτον, η Ευρώπη την την σταθερότητα οικονομική και χρηματική. Αυτά είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά που και τα τρία αφορούν και σχετίζονται με το θέμα της Ελλάδος. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτές τις τρεις διαφορετικές όψεις της Ευρώπης που λαμβάνονται υπόψη και περιέχονται στις 11 Φεβρουαρίου το κείμενο αυτό το οποίο βγήκε σαν συμπέρασμα από την άτυπη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Γι' αυτό και ασχολούμεθα με το πρόβλημα της Ελλάδας μιλώντας για αλληλεγγύη και για την δέσμευσή μας να προχωρήσουμε στην εξασφάλιση σταθερότητας για την Ευρωζώνη. Είμαι βέβαιος ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που είναι το ίδιο αυτό τη 11 η Φεβρουαρίου, αυτό το ίδιο Συμβούλιο πρόκειται να επαναβεβαιώσει την πρόθεση εξασφάλισης της σταθερότητας. Και επομένως θα στείλουμε ένα ισχυρό, αποφασιστικό μήνυμα ότι θέλουμε στήριξη της οικονομίας, στήριξη του ευρωπαϊκού νομίσματος. Φυσικά και αυτό θα γίνει λόγω της αλληλεγγύης και ξέρουμε ότι και κάποιοι ευρωσκεπτικιστές ποθούν την αποτυχία. Όχι, αυτό όμως δεν πρόκειται να γίνει. Αυτό που θα γίνει θα είναι η επιβεβαίωση της πολιτικής βούλησης για αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για αλληλεγγύη στην Ευρωζώνη. Και θα δούμε τι θα γίνει και την επόμενη μέρα. Μεσοπρόθεσμα. Πώς δηλαδή θα βρούμε τη διέξοδο από την κρίση. Για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε σε μια οικονομική ανάκαμψη που αναφέρεται σε αυτό το κείμενο και μιλούμε εδώ και για κάποιους πιο μακρόπνους στόχους. Η οικονομική συνοχή, η εδαφική συνοχή, η κοινωνική συνοχή σε σχέση με το Ταμείο Αλληλεγγύης και άρα χρειαζόμαστε μια διαφορετική υποπτία, διαφορετική από ό,τι πρόβλεπε η Συνδίκη Λισαβόνα. Να τι θα πει πρωτοπορία ευρωπαϊκή. Από του στόχοι που έχει η Συνδίκη Λισαβόνα που δεν είναι η στατική τη Λισαβόνα για απασχόληση, α πούμε, για άλλου κοινωνικού στόχου. Και γι' αυτό χρειάζεται κάποιο παρακολούθηση, έλεγχο, εποπτεία και παρακολούθηση του αν τηρούνται οι στόχοι, πράγματα που δεν τα έχει η στατική. Επίση κάποια κίνητρα ε, σε σχέση με τα διορθωτικά ταμεία. Τίποτα αυτό δεν υπήρχε στην παλιά στρατηγική της Λισαβόνας. Είναι κατακλείδη. Πρόεδρε, να σου πω για αυτό που είπε ο κ. Γκαρθία Μαργάγια. Γιατί ήταν ο μόνος που απευθύνθηκε άμεσα στην ε, Προεδρία την Ισπανική, επικοινωνώντας την. Το Συμβούλιο και η Προεδρία προχωρούν σε στενή συνεργασία και σε συντονισμό επί τη βάση της κοινοτικής μεθόδου με τον πρόεδρο του Συμβουλίου, τον κύριο Φανερόμπαη. Χέρι-χέρι με την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Στενή συνεργασία προς επίτευξη των μεγάλων στόχων. Εσείς αναφερθήκατε στην οικονομική πολιτική, αλλά για πέστε μου, δεν συμφωνείτε ότι Η αποφάσει που λαμβάνει το Συμβουλίο όσον αφορά αυτή τη ε, δέσμευση τη Ευρώπη για την σταθερότητα τη Ευρωζώνης. Αυτό δεν είναι πράξη κατεύθυνση και διεύθυνση και χαλιναγώγηση τη Ευρώπη. Και έτσι προχωρούμε προ τη στρατηγική του 2020. Και ε, τα όσα αποφασίστηκαν συνεκέντρωσαν την συνένεση των περισσότερων πτέρυγων του Κοινοβουλίου. Και τώρα πάμε στην διακυβέρνηση. Και εκεί δεν ισχύει το ίδιο. Για πέστε μας, δεν συμφωνείτε. Και άλλωστε υπάρχει αυτή η πάγια συνεργασία μας με το Κοινοβούλιο όσον αφορά την οικονομική εποπτεία. Και η συνεργασία μας πρόκειται να μας οδηγήσει το συντομότερο σε μια συνεργασία εμάς με εσάς. Και έχουμε και τον οδηγία το ΣΟΣ που επίση και αυτό αποτελεί άλλο ένα λιθαράκι που βάζουμε στην διακυβέρνηση την οικονομική. Πρόκειται για πρόταση που θα κατεβάσει η Κομισιόν για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών για την εφαρμογή του άρθρου 136 της Συνήθισης Λισαβόνα. Επίσης, κρατούμε τα ενία της Ένωσης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βρούμε την έξοδο από το αδιέξοδο του χρέους. Του χρέου μέσα σε αυτή την κρίση μέσα στην κοινωνική πίεση να βγούμε από την κρίση, να βοηθήσουμε τους μη προνομιούχους, τους πιο ευάλωτους. Αυτό θα πει Προεδρία, αυτό θα πει το να κρατάμε το πιδάλιο της Ένωσης και αυτή την εβδομάδα στην πράξη θα πρόκειται να δείξουμε την ελληνική μας προς τον ε, ε, ελληνικό λόγο, προς την ελληνική κυβέρνηση. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Δυστυχώ δεν μπορείτε να μιλήσετε κύριε Γκασία Μαργάγιο με την μπλε κάρτα. Αυτό αφορά μόνο θέματα που αφορούν, που ελέγξαν από βουλευτές. Με την παρέμβαση του Υπουργού ολοκληρώνεται η σχετική συζήτηση.